Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της ε, συνεδρίασης. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Ήδη πόρει ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες ε, των πολιτών ε, και θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στους εκπροσώπους Συμβουλίου και Επιτροπής θα σας πω ότι μπορείτε ηλεκτρονικά να δηλώνετε αν θέλετε το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας της μπλε κάρτας. Έχετε οδηγίες και στο εδρανό σας και έχετε λάβει και ηλεκτρονικά τις σχετικές πληροφορίες. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα και επίσης παράλληλα με το ηλεκτρονικό σύστημα μπορείτε και με το συνηθισμένο τρόπο σηκώνοντας δηλαδή ένα ε, χαρτί ή ενημερώνοντας ε, τις υπηρεσίες της Ολομέλας. Αυτό αυθόρμητα μπορείτε να στήσετε να το λόγο. Επίσης παρακαλώ να έχετε την κάρτα ψηφοφορίας μαζί σας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα και δεν μπορείτε όμως από το γραφείο σας με email να ζητάτε το λόγο, μόνο εδώ προσωπικά, αυτοπροσώπως ή με το ε, σύστημα που σας ε, είπα. Ήδη από τώρα λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα. Και εδώ μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε τις δηλώσεις ακούγοντας καταρχάς την εκπρόσωπο της Φιλανδικής Πρέσης, την κυρία Τουπουράινεν. Honorable Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Επίτροπε, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέσει ακριβώς τα πλαίσια για τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέχρι το 2027 και ο στόχο μας είναι να έχουμε ένα ισορροπημένο πλαίσιο που να καλύπτει και νέε προτεραιότητες αλλά και τις παραδοσιακές μας πολιτικές και να συνεισφέρει στου κοινού ευρωπαϊκού στόχους. Δεν είναι εύκολο βέβαια να πετύχουμε αυτούς τους ουσιαστικούς στόχους, αλλά δουλεύουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Το χρονοδιάγραμμα επίσης είναι και αυτό δύσκολο, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα θεσμικών αλλαγών. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί πάρα πολύ προς αυτό το σκοπό. Η σημερινή συζήτηση πάντως μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ προεδρεύω τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αλλά επίσης εκπροσωπώ και το Συμβούλιο σε όλες τις Ολομέλειες, κάτι το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να συζητώ τακτικά μαζί σας και να σας ενημερώνω. Και στο πνεύμα της καλής διοργανικής ε, συνεργασίας και με το προηγούμενο που έχει θέσει η προηγούμενη Προεδρία και ελπίζουμε και η επόμενη θα ακολουθήσει, θα έχουμε τακτικά ανταλλαγή απόψεων πριν και μετά ε, τις ε, Ολομέλειες, στον ΤΑΚ, όταν θα έχουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο στην ημερήσια διάταξη ω μοναδικό θέμα. Οι προκλήσει είναι πολλέ, λοιπόν και οι προτεραιότητέ μα κοινέ. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θέλει να ανταποκριθεί στι σημερινέ και στι μελλοντικέ προκλήσει, έτσι ώστε να γίνει κατανομή των δαπανών με όσο γίνεται μεγαλύτερη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Οι παραδοσιακές πολιτικές στηρίζονται και διατηρούμε επίσης και υψηλό επίπεδο στην γεωργία στην Ευρώπη. Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα συνεχίσουμε με τις συγκλήσεις για να πετύχουμε μια βιώσιμη γεωργία. Η χρηματοδότηση του αγροτικού κόσμου είναι κάτι πολύ σημαντικό και μία από τις κύριες προκλήσεις της εποχής μας είναι η κλιματική αλλαγή. Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον μας και είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώνεται αν δεν κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Πολλές φωνές ακούγονται, πρώτα απ' όλα της νεολαίας μας, που μας ζητούν να κάνουμε περισσότερα. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο λοιπόν είναι ζωτική σημασία ε, γιατί θα μας οδηγήσει στους ε, στόχους που έχουμε θέσει για το 2030 όσον αφορά το κλίμα. Οι χώρε ε, μέλη φαίνεται να συμφωνούν με το στόχο του 25% ακόμα και αν για μερικέ το 25% είναι το ανώτατο και για άλλε είναι το κατώτατο όριο. Πάντως ο στόχος μας ε, για το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα είναι κάτι που μοιραζόμαστε όλοι και άρα χρειάζεται ένα ταμείο το οποίο να διευκολύνει την δίκαια μετάβαση προς το ουδέτερο αυτό αποτύπωμα άνθρακα. Επίσης θέλουμε καινοτομία, έρευνα που θα στηρίξει το πουδουπού και χρειάζονται βέβαια και μεγάλες αλλαγές στο ψηφιακό κλάδο. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της έρευνας, ε, της ε, ανάπτυξης και της κοινοτομίας. Το μελλοντικό λοιπόν πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να ευθυγραμμίζεται και με νέες προτεραιότητες. Μετανάστευση, Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική προσέγγιση. Χρειάζεται χρηματοδότηση από διάφορους τίτλους του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις διάφορες πτυχές της μετανάστευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συγχρόνω οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Μια από τις μεγαλύτερε χώρες μέλη όπου να είναι φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε με όλους τους υπουργούς και πολλοί έχουν εκφράσει την ε, ανάγκη ο νέος προπολογισμό να αντικατοπτρίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τώρα τους ίδιους πόρους, πρέπει επίσης να προσφέρουν ένα σύστημα δίκαιο με διαφάνεια για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με ελάχιστο βάρος για τις χώρες μέλη. Από πλευράς της Προεδρίας για τους νέους ίδιους πόρους. Η πρόταση όσον αφορά τα πλαστικά και τις συσκευασίες χαίρει της μεγαλύτερης στήριξης από τις χώρες μέλη. Όσον αφορά επίσης τους ίδιους πόρους μας πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι και εδώ χρειάζεται συνένεση μεταξύ όλων των χωρών μελών. Τώρα, Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, το να στηρίζουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε είναι κάτι που ξεκινάει από το σεβασμό του κράτου δικαίου και την προστασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλε τι χώρε μέλη. Το κράτο δικαίου δεν είναι μια πολιτική δήλωση που κάνουμε, αλλά είναι ένα νομικό καθεστώ. Από πλευρά τη Προεδρία, λοιπόν, το άρθρο 2 τη συνθήκη που αναφέρεται στο κράτο δικαίου δεν πρόκειται να ισχύσει από μόνο του και αυτό πρέπει να αντικαταπτρίζεται στην πολιτική μα, στο πολιτικό μα έργο. Το κράτο δικαίου ενιαίο, είναι ζωτική σημασία στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί συμπεριλαμβάνει την πρόταση για την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού από δυναμίε όσον αφορά το κράτο δικαίου. Και είναι μια πρόταση η οποία ισχύει εξίσου για όλε τι χώρε μέλη και για όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπω ισχύει και το κράτο δικαίου εξίσου σε όλε τι χώρε. Το κράτο δικαίου λοιπόν και η δημοκρατία αποτελούν τα θεμέλια τη ελευθερία στην Ευρώπη, τη δημοκρατία τη ευημερία. Η προστασία του συνδέεται επίση με την νομιμότητα και με την καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις προτεραιότητες λοιπόν της Φιλανδικής Προεδρίας είναι να διασφαλίσει την προστασία του κράτους δικαίου και να ενισχύσει την σύνδεσή του με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Μετά τις κατευθυντήριες γραμμές ε, των ε, ηγετών μας θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να έχουμε ένα ισορροπημένο μέσο το οποίο θα βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, γνωρίζω τις ανησυχίες σας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τώρα το έργο της Προεδρίας στο Συμβούλιο έχει προχωρήσει. Έχουμε ακούσει τις χώρες μέλη και τις δικές τους προτεραιότητες. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων να δώσουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές. Προς αυτό το σκοπό η Προεδρία ετοιμάζει ένα έγγραφο το οποίο θα διευκολύνει τις πρώτες συζητήσεις των ηγετών μας στην διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου. Φυσικά εννοείται από τις αντιδράσεις των αντιπροσωπιών και πάνω απ' όλα από τον ίδιο τον ε, πρόεδρο Τάσκ και πώς θέλει να προχωρήσει η συζήτηση αυτή. Και βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών των ε, ηγετών μας θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένα νούμερα ώστε να διευκολυνθεί η απόφαση μέχρι τα τέλη της χρονιάς όπως είπε τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι η Προεδρία έχει δεσμευτεί απόλυτα να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων επί του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι επίσης ζωτική σημασία να συνεργαστούμε μαζί σας και με τις προηγούμενες προεδρίες και να προχωρήσουμε σε τομακές προτάσεις προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση από όλου. Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και προσβλέπω στη συζήτησή μα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τουπουράινεν. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χαν, δεν ε, είδα ότι ο κύριος Ριβέρα ήθελε το λόγο επί της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι ήθελα το λόγο επί της διαδικασίας. Ε, συγγνώμη που γίνεται αυτό στο μέσο της συζήτησης, αλλά χθες έγιναν διάφορα ε, στο πλαίσιο της εκλογής ε, του προεδρίου στην εκπροσωπεία Κάρι Φόρουμ μια σε πρόσωπος από τη δική μας ομάδα η ΝΤΕ είχε οριστεί στις 17 Ιουλίου στην αντιπροσωπεία Κάρι Φόρουμ είναι τακτικό μέλος αυτής ε, της αντιπροσωπείας από τον Ιούλιο. Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας κοινοποίησε ότι δεν μπορούσε να ε, κατέλθει ε, υποψήφια διότι δεν είναι μέλος της αντιπροσωπείας Κάρι Φόρουμ. Είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση της πρώτης αντιπροέδρου με βάση τους κανόνες δεών που βέβαια δεν γίνονται σεβαστοί αλλά τέλος πάντων. Πάντως δεν μπόρεσε να υποβάλει υποψηφιότητα και επειδή Έχουμε ακούσει κάποια ανησυχητικά ε, λόγια για ένα είδος αποκλεισμού, το λεγόμενο κορδόν σανιτέρ, ε, που δεν μας επιτρέπει να πάρουμε ε, κάποια αξιώματα. Δείχνει όλο αυτό ότι υπάρχει βούληση να μπαίνουν στο περιθώριο τα μέλη της ομάδας ID. E ID. Ή, αν δεν ισχύει αυτό, έγινε κάποιο παρόραμα ή κάποιο σφάλμα. Θα ήθελα λοιπόν να διορθωθεί αυτό για να μπορέσει υποψήφιο άμα μας ε, να πάρει αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Για να δω ποιος θέλει το λόγο. Μαριάννη, για το ίδιο θέμα θέλετε το λόγο. Όχι. Τότε να περιμένετε σας παρακαλώ, ο κύριος Βίλαντ. Ναι, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Για τον κύριο Ριβιέρα να πω δεν ε, είναι χωρίς λόγο που ψηφίζουν οι αντιπροσωπείες. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων που αποφασίζουν ε, και σίγουρα λαμβάνονται υπόψη και πολιτικές σταθμίσεις και παράμετροι ε, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, μπορεί φυσικά οποιοδήποτε να θέσει την υποψηφιότητα αφού είναι τακτικό μέλος και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο ε, θα σας ε, ενημερώσω, θα δω γιατί το πρώτο είναι ένα τυπικό το οποίο προβλέπεται από τον ε, εσωτερικό κανονισμό ότι ένα τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Το αν όμως θα εκλεγεί ή όχι στη θέση για την οποία έχει θέσει υποψηφιότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μαριάννη το έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να παρέμβω όσον αφορά το σύστημα DONT και αυτά που έγιναν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε 13 κανονικέ ε, εκθέσει για την πεντετία τη για 13 χώρε που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με συμφωνίε γειτονία είτε προενταξιακά. Αυτέ οι 13 εκθέσει λοιπόν καταναμήθηκαν μεταξύ τριών πολιτικών μονάδων μόνο Σιέρι, Γκουε και το ΙΝΤΕ αποκλείστηκαν πλήρω. Και μα εξηγούν ότι οι εκθέσει αυτέ δεν υπολογίζονται βάσει του κανόνα DONT. Μα κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε πότε εφαρμόζεται αυτό ο κανόνα DONT και πότε όχι. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε διακρίσει. Με τι 13 εκθέσει θα μπορούσαμε κάπω αναλογικά να τι κατανείμουμε, δεν νομίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Μαριάννη. Η απάντησή μου αφορά ε, εδώ ε, την, ε, και αυτό που είπα για τον κύριο συνάδελφο και το δεύτερο τμήμα της παρέμβασή του φυσικά ε, και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και υπάρχει ε, η πολιτική ομάδα, η μάλλον πολιτικές ομάδες και αυτές λαμβάνουν απόφαση. Δεν ε, μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Η επιλογή των θέσεων είναι κάτι τελείω διαφορετικό καθώς και η απόνομη των εκθέσεων. Ο κύριος Χάνιχ τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το νέο ΠΔΠ. Ξέρω ότι είναι στρατηγική σημασία ε, το ζήτημα αυτό, καθότι θα διαμορφώσει το μέλλον ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη δεκαετία και αναγνωρίζω το πολύ σημαντικό εντατικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίω των ε, συνεισηγητών και τη διαπραγματευτική ομάδα που είναι οι κύριοι Μάρκε Χέρε και Σάντρε Φερναντέ και σίγουρα ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει υπόψη όλα αυτά. Υπάρχει και η ανταλλαγή απόψεων την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και φυσικά ενθαρρύνω τη Φιλανδική Προεδρία να λάβει υπόψη τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδιάμεση έκθεση που ενέκρινε τον Νοέμβριο τη περσινή χρονιά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μια σημαντική συνεισφορά στι διαπραγματεύσει για το προσεχέ πιδελταπή ένα χρόνο μετά και μετά τι ευρωεκλογέ του Μαΐου. Ήταν σημαντικό να μην υπάρχει καμία απολύτω ασάφεια σε ό,τι αφορά ε, τη σταθερή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό χαιρετίζω το ότι στο ψήφισμα αυτό οι θέσει ε, του 2018 γίνονται δεκτέ στο μεγαλύτερο μέρο του και λαμβάνω υπόψη και τα νέα στοιχεία του πολιτικού αυτού ψηφίσματο, τα οποία θα ε, τα σχολιάσω στη συνέχεια. Αλλά καταρχά θα ήθελα να σα υπενθυμίσω τη θέση σε σχέση με το συνολικό επίπεδο των δαπανών. Είναι ένα από τα ζητήματα, ίσω το σημαντικότερο ζήτημα ε, των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει σε ό,τι αφορά τον επόμενο προπολογισμό να έχουμε το 1 τρίτο του ακαθάριστου εθνικού ε, ευρωπαϊκού εισοδήματο. Και πολλά κράτη-μέλη 1,3%. Και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ε, δυνατότητα καλυφθούν οι αποκλήσεις που υπάρχουν μεταξύ ε, των θέσεων Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε ε, όσο το δυνατόν δε συντομότερα για τον μελλοντικό μακροχρόνιο προϋπολογισμό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ένωση καλείται να κάνει περισσότερα ε, σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε και με καλύτερο τρόπο. Ο προπολογισμό πρέπει να εστιάσει στην ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Περισσότεροι πόροι ε, πρέπει να δοθούν για προγράμματα που άπτονται τη έρευνα καινοτομία, κλιματική αλλαγή, ψηφιακή, τεχνολογία, ασφάλεια, διαχείριση νόρου κτλ. Βέβαια δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή μα και με την πραγματικότητα. Ε, η εξοικονομήσεις ε, στη κοινή γεωργική πολιτική, την πολιτική συνοχή είναι αναπόφευκτες και υπάρχουν αυτοί οι δύο περιορισμοί. Γι' αυτό και προτείνουμε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 1,14 για ε, το ε, σε σχέση με το ΑΕΠ και νομίζουμε ότι αυτό είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση Δεχόμαστε τις περισσότερες θέσεις του Κοινοβουλίου της περσινής χρονιάς. Αλλά υπάρχουν και κάποια νέα στοιχεία σε αυτό το πολιτικό ψήφισμα. Ε, το πρώτο είναι η χρηματοδότηση των πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών τη εκλεγής σα Προέδρου τη Κομισιόν, όπω καταλαβαίνετε δεν μπορούν να ε, παραβιάζουν τι προνομίε ε, τη επόμενη ε, επιτροπή και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ήδη έχουμε ένα πλαίσιο ε, πολύ σταθερό για αυτές τις προτεραιότητες. Έχουμε το δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης που είναι ένα στοιχείο. Το άλλο είναι το κράτος δικαίου που αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα ε, του μακροπρόθεσμου προπολογισμού. 120 δις ε, για εξωτερικές επενδύσεις και πιο στενή εταιρική σχέση με την Αφρική. Ενίσχυση επίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 22 φορές περισσότερος ο προ... μεγαλύτερος ο προϋπολογισμός δηλαδή από 590 εκατομμύρια περνάει σε 13 δις και σίγουρα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με ταχύτητα, με αποφασιστικότητα ώστε οι πολιτικές κατευθυντές γραμμές της εκλεγής της Πρόεδρου να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δράσεις και να πλαισιωθούν από αυτή τη συμφωνία. Δεν θα πρέπει να έχουμε επιζήμιες καθυστερήσεις για τη δρομολόγηση των προγραμμάτων. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των περιφερειών, προς όφελος ερευνητών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών, νέων κτλ. Έρχομαι τώρα στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ποσοτικοποιημένους και πιο φιλόδοξους στόχους ε, για τις δαπάνες σε σχέση με το κλίμα. Θέλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας στο Παρισί για την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να πρωτοστατούμε, να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και θέλουμε υψηλότερους στόχους. Το 25% του πιδελταπή γύρω στα 320 δις. Θέλουμε να ε, ανατεθούν αυτά τα κονδύλια για κλιματικά προγράμματα αξιόπιστο αυτό ο στόχος, ε, πιστεύουμε και εφικτός αυτό το 25%. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με κάθε πρόγραμμα και πώς μπορεί να συνεισφέρει στην κλιματική δράση. Κάποια προγράμματα θα συνεισφέρουν σημαντικά στην κλιματική δράση, κάποια άλλα μεταξύ άλλων και αυτά για τα οποία προτείνεται ενίσχυση όπως ε, Ενέα Αγορά, Erasmus, ε, Creative Europe. Δημιουργική Ευρώπη, ΕΣΕΦ, δεν θα ε, συνεισφέρουν τόσο. Αν θέλετε να υπερβούμε το 25% θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Παραδείγματος χάρη, κλιματικοί στόχοι προγραμμάτων που ήδη συνεισφέρουν στην κλιματική δράση θα πρέπει να αυξηθούν. Άρα Πολύ ψηλότεροι θα πρέπει να είναι οι στόχοι, παραδείγματο για την κοινωνική πολιτική, για το ΕΤΠΑ, για το Ταμείο Συνοχή λόγω της ε, κρίσιμη μάζα του στον προπολογισμό ή θα μπορούσαν ε, σε σχετικού όρου να μειωθούν ε, τα κονδύλια που δίνονται σε προγράμματα που δεν συνεισφέρουν στην κλιματική δράση. Και αυτό θα επηρέαζε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλες νέες προτεραιότητε όπω το Εράσμου, η Άμυνα, η Ασφάλεια η, διατήρηση το, διαχείριση των συνόρων. Ε, Επομένω, οι μαθηματικέ επιλογέ είναι αυτέ. Ε, σίγουρα είναι σκληρέ οι επιλογέ. Ε, θα ασκηθούν σίγουρα τα δικαιώματα και θα μπορέσουν να κάνουν τις προτάσεις τους και τα κράτη-μέλη. Δεν έχει άλλωστε το Συμβούλιο ακόμη καταλήξει σε μια θέση ότι αυτό το πει. Εμεί ω Κομισιόν θα διευκολύνουμε το διάλογο, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε σε Συμβούλιο και σε ε, Κοινοβούλιο τεχνικέ πληροφορίε για διαφάνεια, ανοιχτό πνεύμα, επικοδομητική συνεργασία. Τέλο, το ψήφισμα ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη ε, το αργότερο στι αρχέ του 2020, ώστε να υπάρχει συνέχεια στη χρηματοδότηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίε και να συμφωνηθεί το νέο πι. Όπως πολύ σωστά λέτε, η συνθήκη στο άρθρο 312 και ο κανονισμός πι παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την περίπτωση που δεν θα έχει υπάρξει συμφωνία. Δεν είναι λοιπόν τώρα ε, η ώρα να σκεφτούμε πρόσθετα μέτρα, γιατί προ το παρόν προτεραιότητά μα ε, είναι εγκαίρα να πετύχουμε συμφωνία για το νέο ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τι σχετικέ τομεακέ πράξει. Σα ευχαριστώ για την στεναρή σα υποστήριξη και για τη μεταρρύθμιση του συστήματο των ιδιών πόρων. Να υπάρχει ευελιξία στο πιδελταπή και να θεσπιστεί ένα μηχανισμό για την προστασία του ενωσιακού προπολογισμού σε περίπτωση γενικευμένων ε, προβλημάτων στον τομέα του κράτου δικαίου. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, συμφωνώ μαζί σα ότι είναι καιρό πλέον να, να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε των πολιτών. Έχουμε συλλογική ευθύνη όλοι μας να συμφωνήσουμε για τον μακροπόθεσμο προπολογισμό της Ένωση έγκαιρα, ώστε οι νέε γενιέ προγραμμάτων να μπορέσουν να ε, ε, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στις δηλώσεις των συναδέλφων. Ο κύριος Όλμπριχτ είναι ο πρώτος ομιλητής ε, για 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, αυτή είναι η αλήθεια. Ο χρόνος περνάει γρήγορα τα πανεπιστήμια, οι ε, κοινότητες, ε, οι φοιτητές που θέλουν να φύγουν για το Εράσμος περιμένουν τα αποτελέσματα για τον προπολογισμό μετά το 2020. Θα υπάρχει προπολογισμό ή δεν θα υπάρχει. Πότε θα ληφθεί η απόφαση, πότε θα ληφθούν γενικότερα οι αποφάσεις. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε με την γενική έκθεση με τις διάφορες εκδοχές και παρουσίασε τις θέσεις της το Μάιο του 2018. Ενάμιση χρόνο μετά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, απάντησε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν παρά το γεγονός ότι η διαδικασία όπως προβλέπεται από τις συνθήκες δεν προβλέπει τέτοια υποχρέωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο όμως ε, με αίσθηση ευθύνη υπέβαλε την πρότασή του και τη θέση του το Νοέμβριο. Η θέση αυτή είναι καθόλου ρεαλιστική. Έχουμε λάβει υπόψη τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν επινοήσαμε πράγματα εκ νέου. Απλώς ε, δώσαμε την έγκρισή μα για κάποιες νέες προτεραιότητες. Ε, ε, αποφασίσαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ορίζοντα 2020 και κυρίω πρέπει να ενισχύσουμε και το Εράσμους. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική μα ε, θέση. Πιστεύουμε επίση ότι οι λεγόμενε παραδοσιακέ πολιτικέ δεν μπορούν αυτομάτως να υποστούν μειώσεις. Ποιο θα είναι το κόστος του Brexit. Το Κοινοβούλιο σήμερα λέει ότι ο χρόνος περνάει και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα προπολογισμό και δεν θα χρειαστούμε μόνο κάποιες συναντήσεις μαζί σας ε, για ανταλλαγή ε, κολακιών. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για να δώσουμε και την έγκρισή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μάρκες. Έχει το λόγο τώρα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ του Περχάινεν, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, να σας υπενθυμίσω τον τίτλο αυτής της συζήτησης ώρα να ικανοποιηθούν οι προστοκίες των πολιτών. Γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ. Πρέπει να εγκρίνουμε τον προπολογισμό στο ύψο των δεσμεύσεων και των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, επιβεβαιώνουμε τη θέση της έκθεσης του Δεκεμβρίου του 2018, αλλά αυτή τη στιγμή και μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Επικαιροποιούμε την ε, εντολή διαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη και το αποτέλεσμα των ευρωκλογών που διεξήχθησαν το Μάιο το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να καθοριστεί με 1,3% ακαθόριστο εγχώριο εισόδημα. μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πρικοδοτήσουμε παρκώς ε, τη μεταναστευτική πολιτική, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας και να υπάρχει ένας ισχυρός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και την κατάλληλη ΚΑΠ. Υπάρχουν και τα θέματα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, τα οποία πρέπει να είναι οριζόντια. Πρέπει να έχουμε μια ουδέτερη οικονομία σε θέματα άνθρακα και χρειαζόμαστε κοινωνικές ε, διατάξεις για να μην αποκλείεται κανείς. Ε, πρέπει να υπάρξει ένας νέος μηχανισμός προκειμένου να ε, γίνεται και περικοπή των κονδυλίων σε χώρες που δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου οι ε, επιπλέον πρωτοβουλίες και οι δεσμεύσεις της κυρίας Φοντερ θα πρέπει να δούμε και πώς θα προχωρήσουν. Αλλά για να έχουμε νέες ε, πρωτοβουλίες πρέπει να υπάρχει και κατάλληλα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Και αυτά θα πρέπει να έρθουν επιπλέον. Για παράδειγμα για το ε, περιβόητο Green Deal. Ε, είμαστε ικανομένοι από τις προτάσεις της κυρίας Φοντερ να υπάρξουν νέες προτάσεις νομοθεσίες για να έχουμε ένα νέο κατάλληλο ιδίων πόρων. αυτό που μας κάνει όμως να αναρωτήσουμε αναρωτιόμαστε είναι αν θα αλλάξει τώρα ο τρόπος χρηματοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις ε, βασικές ε, πολιτικές προτεραιότητες. Θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να συνάδουν και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το θέμα των ιδίων πόρων. Θα πρέπει Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε και τις ε, τομεακές πτυχές ε, και να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωση και να δούμε επίσης και τι θα γίνει με την πρόταση για το κράτος δικαίου. Χρειαζόμαστε ένα ε, σαφές πλαίσιο ώστε να μην υπάρξει και κενό μεταξύ του τέλους του προηγούμενου PDP και τη έναρξη του νέου. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Μάρκε. Τώρα δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Αγέ. Ευχαριστώ, Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, σίγουρα θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τι συζητήσει στο Συμβούλιο. Γιατί ανυπομονεί το Κοινοβούλιο. Πριν από 17 μήνε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή τη για το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε αμέσω να εργάζεται και εξέφρασε την θέση του και τι προτεραιότητέ του. Περιμένουμε από τότε να προχωρήσει το Συμβούλιο σε διάφορα ζητήματα και πιέζει ο χρόνο. Επιτέλου πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα στι διαπραγματεύσει. Επίση ήρθε η ώρα να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Η γραμμή που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφή και σήμερα επιβεβαιώνουμε τι προτεραιότητέ μα. Διατήρηση του προπολογισμού για την κοινή γεωργική πολιτική πολιτική για τη συνοχή, την ενίσχυση των εμβληματικών προγραμμάτων όπω είναι το έρασμο και άλλα, νέε πιστώσει για νέε προκλήσει ή ακόμα και δημιουργία ενό μηχανισμού που συνδέεται με το κράτο δικαίου. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να ανταποκρίνεται και στι ανάγκε για την κλιματική αλλαγή και την βιοπικιλότητα. Για τα θέματα αυτά, η εκλεγμένη πρόεδρο Βοντερ Λάιεν είπε ότι θα υπάρξει ένα New Deal και ότι θα υπάρξει και φόρο για τον άνθρακα στα σύνορα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι πρωτοβουλίε. που χαιρετίζουμε, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα ε, δημοσιονομικά ε, πλαίσια, από τα κατάλληλα κονδύλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λένε θέλει όλο να ξοδεύει περισσότερα. Όχι, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Αν έχουμε τέτοια κονδύλια και θέλουμε περισσότερε πρωτοβουλίε, πώ θα γίνει. Κάπου θα γίνουν αλλού περικοπέ. Οπότε θα έχουμε λιγότερο αποτελεσματικέ δημόσιε πολιτικέ. Όχι, μην ε, δίνουμε τροφή στου ευρωσκεπτικιστέ. Το σύστημα τώρα των εσόδων που το έχουμε από το 1970 έχει ξεπεραστεί. Σήμερα οι εθνικές συνεισφορές ε, τροφοδοτούν τη λογική των δίκαιων επιστροφών. Εμείς διατηρούμε ένα σύστημα όπου τελικά έχουμε τις εθνικές προσεγγίσεις ενώ πρέπει να δώσουμε περισσότερη αξία στην προστιθέμενη ακριβώ ευρωπαϊκή αξία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με το νέο πλαίσιο χωρίς νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε ότι τώρα το μπαλάκι είναι στο δικό σα το γήπεδο. Γνωρίζετε ποιε είναι οι θέσει μα. Εμεί περιμένουμε τι δικέ σα, ώστε να προχωρήσουν επιτέλου οι συζητήσει προ το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων σα ευχαριστούμε κύριε Χάιερ. Τώρα για δυόμιση λεπτά το λόγο έχει ο συνάδελφο Αντρέσεν. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση με το κλίμα, κοινωνική διάσπαση, ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντικά ζητήματα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε με εθνικό τρόπο πλέον. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί πράσινοι θέλουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να προσφέρει μέλλον ε, στου νέου και να είναι ουδέτερο προ το κλίμα μέσα σε 20 χρόνια. Και αυτό πρέπει να κάνουμε επενδύσει. Ε, το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ μα προσφέρει τώρα την ευκαιρία γι' αυτό. Και θέλω να πω ευθύ εξ αρχή πω η θέση τη Ομοσπονδιακή ε, Κυβέρνηση τη Γερμανία και άλλων κρατών βλάπτει την Ευρώπη. Διότι το 1% ε, του ΑΕΠ για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον αγώνα κατά του κλίματο δεν επαρκεί. Είναι ελάχιστο αυτό το ποσοστό. Και η Άγγελα Μέρκελ και ο Όλαφ Σόλτ, Υπουργό Οικονομικών, πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο σθένος. Ε, δεν θα πρέπει να βάζουν φρένο ε, σε όλα αυτά και πρέπει να αλλάξει θέση διότι εάν κόψουμε τον προϋπολογισμό περιορίζουμε τη δράση για το κλίμα λίγα για την έρευνα θα δαπανώνται λίγα για το έρασμο θα επενδύονται και βέβαια έχουμε και κάποιες εισαγγελικές επιδοτήσεις ε, για μέτρα που βλάπτουν ε, το κλίμα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να προωθήσουμε σίγουρα μια βιώσιμη γεωργία και την οτροφία. Επίσης ε, θέλουμε να επενδύσουμε και στην βελτίωση του συνδρομικού δικτύου. Η βελτίωση των οποδομών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας τους πρασίνους. Βλέπουμε πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν ε, σε πολύ ε, άσχημες συνθήκες φτώχειας και πρέπει τη φτώχεια αυτή να την καταπολεμήσουμε. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο η φτώχεια στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν ε, να σας πούμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό ε, πάνω σε αυτό το πι. Θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να δράσουμε και στις ε, διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε σκληροί, διότι εδώ μιλάμε για το μέλλον μας. Μιλάμε για το μέλλον όλων των Ευρωπαίων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Άντρεση. Για δύο λεπτά ο κύριος Τζάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες ε, από τότε που εδώ στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συζητάμε το επόμενο πι, αλλά η πρόοδο κατά την άποψή μου είναι ανεπαρκής και μέχρι και σήμερα παρά τις δεσμεύσεις της Φιλανδικής Προεδρίας ότι θα ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει χώρος για συμφωνία. Αυτό κατά την άποψή μου κυρίως διότι δεν εξετάζεται το επόμενο πι με ρεαλισμό και γιατί η πλειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία προσέγγιση η οποία είναι παντελώς ουτοπική για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το επόμενο ΠΔΠ. Ζητάμε πολλούς πόρους επιπλέον, 200 δις ευρώ επιπλέον για να χρηματοδοτήσουμε κάποια προγράμματα και κάποιες νέες προτεραιότητες. Εγώ όμω φρονώ ότι προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα πρέπει να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό και να θέσουμε την εξή ερώτηση. Αν κάθε φορά που πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ζητάμε περαιτέρω πόρου και τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να του διαθέσουν, κάποιο λόγο θα υπάρχει. Αν είναι καλή μια εγώ πιστεύω ότι οι χρηματοδότες ε, ε, με ικανοποίηση θα διαθέσουν περισσότερα κονδύλια. Αν δεν θέλουν να τα διαθέσουν, είναι σχετικά προφανή ο λόγος ότι δεν θεωρούν δηλαδή αυτά τα προγράμματα και αυτές τις γραμμές ε, δαπανών αποτελεσματικά για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Και εμένα με αποσχολεί το εξή ότι η επόμενη πρόταση για το ΠΔΠ είναι γεμάτη ερεσιμότητες. Ερεσιμότητε, οι οποίε ουσιαστικά θα κάνουν αυτό το εργαλείο αντιδημοκρατικό και οι αποφάσει για τι δαπάνε και την κατανομή των κονδυλίων θα είναι έρμεο κάποιων γραφειοκρατών στι Βρυξέλλες. Ένα τελευταίο πράγμα για του ίδιου πόρου. Ε, να αρχίσουμε να του λέμε με το όνομά του. Οι ίδιοι πόροι είναι νέοι φόροι, παράνομοι φόροι που οι Βρυξέλλες θέλουν να επιβάλλουν στου ευρωπαίου πολίτε. Αυτή δεν είναι η σωστή προσέγγιση και νομίζω ότι σε αυτή την άγουσα θα βρούμε ποτέ την κατάλληλη συμφωνία ώστε το εργαλείο αυτό να είναι στην υπηρεσία των πολιτών και όχι ένα ε, μέτρο πολιτικού εκβιασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσάν. 1,5 λεπτό κύριε Σίλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για ένα ε, ψήφισμα το οποίο καταθέσαμε και η σημερινή συζήτηση λέει ότι είναι ώρα να ικανοποιηθούν προσδοκίες των πολιτών. Κάποιοι λένε ότι ο προπολογισμό πρέπει να μειωθεί, κάποιοι λένε ότι ο πρέπει να αυξηθεί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οδήγησε σε απογοήτευση της χώρες της συνοχής και δεν έχει ληφθεί επαρκώς και το Brexit, ε, διότι ε, η συνοχή θα χάσει πολύ περισσότερα Πρέπει να δούμε επίσης την κατάσταση που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη που μπορεί να έχουν ε, διαφορετικούς προϋπολογισμούς ή ε, διαφορετική γεωργική ανάπτυξη. Τα λοιπάσματα όμως παντού κοστίζουν το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν και εκείνη η γεωργική πολιτική ε, να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στις προτάσεις κομισιών. Δεν μπορούμε να μειώνουμε συνεχώς δαπάνες. Και σε ό,τι αφορά την έρευνα, την επιστήμη, Από πού θα βρεθούν κονδύλια, πού θα έχουμε αύξηση και πού θα έχουμε μείωση. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ανεπαρκή τις προτάσει τη Κομισιόν για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και απαράδεκτε τι περικοπέ που προτείνει ακόμη και στην ισχνή πρόταση τη Κομισιόν το Συμβούλιο όπως θεωρούμε και επικίνδυνη την καθυστέρηση και τη δυστοκία στο Συμβούλιο που επί 1,5 χρόνο έχει ένα φάκελο και δεν τον προχωρά. Ενώ το Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει στο ακέραιο την ευθύνη του. Θεωρούμε ανεπαρκή την πρόταση της Κομισιόν και απαράδεκτη τη στάση του Συμβουλίου, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το ύψος του προϋπολογισμού, όπου το κοινοβούλιο ζητά έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση να ενισχύσουμε την κοινωνική ατζέντα την απασχόληση τη στροφή από τη λιτότητα σε μια βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και όσον αφορά την εσωτερική κατανομή αυτών των κονδυλίων γιατί είναι προκλητικό άδικο παράλογο να πολλαπλασιάσουμε όπως ομολόγησε ο κύριος χαν 22 φορές τις δαπάνες για την άμυνα και να περικόπτουμε τις δαπάνες για την κοινή αγροτική πολιτική και τη συνοχή και να μην δίνουμε τα χρήματα που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδημούλη. Ένα λεπτό κύριο Στάις. Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν πρέπει να πηγαίνει στην άμυνα. Όμως, σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στην άμυνα με 22% αύξηση στο κονδύλιο το σχετικό. Ε, οι χώρες μέλη συνεισφέρουν επίση σε διάφορε διευκολύνσει υπέρ τη ειρήνη, στην ΠΕΣΚΟ και σε ε, οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την άμυνα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να δημιουργήσει έναν Ευρωπαϊκό στρατό. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με αυτόν τον στρατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά ωφέλη από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν για την άμυνα, μόνο έξι χώρες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους του 2% του ΑΕΠ του συνεισφορά στο ΝΑΤΟ η Γερμανία και η Ιταλία δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στι υποχρεώσεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ. Γιατί λοιπόν το ΝΑΤΟ να έρθει και να τους βοηθήσει αν το χρειάζονται τη στιγμή που δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάις. 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο. Εμείς περιμένουμε για άλλη μια φορά το Συμβούλιο. Περιμένουμε ξανά το Συμβούλιο, το οποίο καθυστερεί. Ο πρόεδρος του... Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου δεν ακούει το Κοινοβούλιο και από ό,τι έχουμε ακούσει δεν υπάρχει σεβασμός τελικά απέναντι στους ίδιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτική συνοχή, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε ε, την πολιτική αλίας και συγχρόνως θέλουμε να ενισχύσουμε την έρευνα, την καινοτομία, ε, να στηρίξουμε το κλίμα, τους νέους, το έρασμος, ε, πράγματα τα οποία κανονικά λέει και το Συμβούλιο ότι τα θέλει. 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Όμως, τελικά θα συμφωνήσουμε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μόνο στην περίπτωση που έχουμε και ευρεία συμφωνία για νέους ίδιους πόρους. Οι νέοι ίδιοι πόροι πρέπει να έρθουν με διαφάνεια, με απλοποίηση και θα πρέπει επίσης να εξετάζουν και εθνικές διορθώσεις. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι. Λέει η Επιτροπή ότι χάνεται ένα δισεκατομμύριο στην φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ναι λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα προπολογισμό ο οποίος θα είναι φιλόδοξος, έναν προπολογισμό όπως αυτός που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ενώ το Συμβούλιο τον απορρίπτει. Η Επιτροπή ελπίζει και εμείς επίσης ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες. 1,5 λεπτό το λόγο η κυρία Γκαρδιά Θάμπαλ Ρουμπιάλ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ, σήμερα συζητάμε το ψήφισμα αυτό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει περισσότερη σημασία από ποτέ ακούγοντας αυτά που μας στάνουν από το Συμβούλιο. Πριν από ένα χρόνο εμείς είχαμε τη θέση μας ξεκάθαρη για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βάσει των αναγκών, των προτεραιοτήτων μας, των πολιτικών μας υποχρεώσεων και υπήρχε και ποσοτική έκφραση, δηλαδή με νούμερα πόσο θα έπρεπε να είναι αυτός ο προπολογισμό εξού και το 1,3%. Υιοθετήσαμε επίση μια ξεκάθαρη θέση λέγοντα ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μπορεί να εξαρτάται περίπου αποκλειστικά από τι εισφορέ των χωρών μελών και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο σύστημα χρηματοδότηση που να βασίζεται στην εσωτερική αγορά, σε δίκαια, αφορολογία ε, και στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Με το ψήφισμα αυτό, τέσσερα θέματα βάζουμε. Το ένα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την θέση του του 2018 Δεύτερον, ότι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή απαιτεί μεγαλύτερε υποχρεώσει από αυτέ που αναλάβαμε πέρσι. Τρίτον, ότι η εκλεγμένη πρόεδρο Φοντερ Λάιεν και πολλοί από του επιτρόπους που ακούσαμε ε, στι ακρόασει δεσμεύτηκαν ε, ενωπιών μα να αναλάβουν νέε πρωτοβουλίε οι οποίε δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και γι' αυτό θέλουμε αναθεώρηση. Και τέλο, και το έχουμε πει όλοι, θέλουμε ε, να ξέρετε το εξή. Ένα χρόνο και παραπάνω περιμένουμε το Συμβούλιο. Εμεί δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία μόνο και μόνο επειδή ο χρόνο τρέχει και δεν προλαβαίνουμε. Ναι, μεταβατικά μέτρα. Ξέρουμε ότι η συνθήκη τα προβλέπει. Αλλά βέβαια στην πράξη είναι πολύ πιο περίπλοκο. Οπότε α προσπαθήσουμε να εργαστούμε για να τα καταφέρουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκαρθία Θάμπελ Ρουμπιάλ. κύριο Κέρνερ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κυρίε και κύριοι. Είναι η πρώτη μου ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι εισηγητή ε, τη Ρηνιού για το πολιτέ μεσονομικό πλαίσιο και χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνω το λόγο. Γιατί με αυτό το προπολογισμό θα βάλουμε τα λιθαριά, τους δομικούς λίθους ε, για τον προπολογισμό των επόμενων ετών στο μέλλον και για το μέλλον. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Πρέπει να φέρει πραγματική προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία αυτός ο προπολογισμό και χρειαζόμαστε για τα μείζωνα ζητήματα μεγάλο προπολογισμό και για τα λιγότερο, για τα πιο ελάσσονα, έναν πιο ε, περιορισμένο προπολογισμό. Πρέπει να γίνει δηλαδή σωστή εράργηση ε, προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση, η έρευνα, το εράσμους ε, καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, ε, καταπολέμηση τη τρομοκρατία και προστασία εξωτερικών συνόρων. Στι διαπραγματεύσει ε, όμω, η δική μου ομάδα θέλει να τονίσει το εξή. Ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, να τα λαμβάνουν κάποιοι αλλά να καταπατούν με χέρια και πόδια ε, τις ευρωπαϊκές αξίες. Είμαστε μια κοινότητα αξιών και όποιος δεν υποστηρίζει αυτές τις αξίες θα πρέπει να, πρέπει να παίρνει και κονδύλια. Εμείς από την ομάδα Renew Europe δεν θέλουμε εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τις αξίες, θεμελιώδες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θέλουμε να το τονίζουμε στι διαπραγματεύσει. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτή η πτυχή στι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ και στον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό, κύριο Κογμό. Bonjour, merci. Καλημέρα, ευχαριστώ το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστική σημασία για το κλίμα. Η Ευρώπη έχει ιστορική ευθύνη και πρέπει να υπάρχει προπολογισμό στο ύψο των προκλήσεων. Το κείμενο το οποίο μα υποβάλλεται σήμερα το πρωί έχει κάποιε προόδου. Ε, η ρητή αναφορά στη σεβασμό των στόχων των Παρισίων για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 είναι ε, ένα σωστό στόχο. Αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα. Πώ μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν υπάρχει τίποτα εγγεγραμμένο στο επόμενο ΠΔΠ. Αυτή λοιπόν είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε. Είναι καλό νέο το γεγονός ότι το ε, ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει το ΠΙΔΕΛΤΑΠΟ ε, πει αν, εγκριθεί, αν ενισχυθεί το τμήμα των ιδίων πόρων και πρέπει να κάνουμε περισσότερο για το κλίμα. Πρέπει να έχουμε και ε, φόρο για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ στην κεροζίνη το συντομότερο δυνατόν. Χρειάζεται μια νέα συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Για τα δύο ευρώ που θα λαμβάνονται από τα φόρο αυτό που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να λάβουν, το ένα θα βγαίνει από τον δημόσιο κορβανά και το άλλο θα μένει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να υποστηρίξει τι πράσινε τι πολιτικέ που χρειαζόμαστε. Ο προπολογισμό πρέπει να είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτικών που θα σέβονται τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Κόγμα. Επόμενη η κυρία Λαπόχτα, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάζοντα την πρόταση κοινού ψηφίσματο, κατάλαβα γρήγορα ότι τα πάντα είναι πρόσχημα για να αυξηθεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία, το Common Mars ε, και το, οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν πάντα να. Ε, υποστηρίξουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία αύξηση χωρί προηγούμενο του προπολογισμού που θα επιβαρύνει τον γαλλικό προπολογισμό. Ζητάτε ε, τα 1,324 δι. ένα προπολογισμό ε, τεράστιο. Ε, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλήρη ανικανότητα ενό γραφειοκρατικού οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον προπολογισμό του, να μην θέλουμε δηλαδή να γυρίσουμε προ τα πίσω. Το θέμα είναι ποιο θα υποφαληθεί από αυτή τη νέα χρηματοδότηση. Οι γεωργοί, οι επιχειρηματίε μα, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε υπόκεινται τον αθέμητο ανταγωνισμό από τον πολλαπλασιασμό των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, σίγουρα όχι. Διάβασα το κείμενό σα. Αυτά οι επιπλέον πόροι είναι για να αντιμετωπίσουμε ε, τις νέες ευθύνε σε θέματα μετανάστευση εξωτερικών σχέσεων και άμυνας. Από αυτό το κείμενο ε, ως σχόλιο δεν θα κάνουμε τίποτα. Ε, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους ίδιους πόρους εσόδων και εκεί δίνεται μεγάλη φαντασία. Για παράδειγμα, ε, δικαιώματα στα τελωνία για τα κράτη-μέλη ή κάποια έσοδα τα οποία θα προκύψουν από πρόστιμα και από τιμωρία τιμωρίες και ε, για ε, φόρους για τα πλαστικά. Εγώ ε, στην αντιπροσωπεία μου θεωρώ ότι θα πρέπει καταρχάς να μειώσουμε το προηγούμενο πι στο ε, 2021 και κόβει ο Πρόεδρος στην ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαπότ. Ένα λεπτό ο κύριος Σόντσα. Ευχαριστώ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση το νέο PDP. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά διαπραγματεύσει όσον αφορά τι δαπάνε αλλά και όσον αφορά του πόρου. Θα θέλαμε να πρόκειται για ένα προπολογισμό που βασίζεται στα πραγματικά προβλήματα και οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να πετύχουμε μια στέρεα συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να παρατείνει το σημερινό πουδουπού για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αν μη τι άλλο τους Ευρωπαίους δικαιούχους. Ένα τέτοιο κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι διαπραγματεύσεις επίσης να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει και πρόταση για νέου ίδιου πόρους. Εγώ υπενθυμίζω ότι κάθε νέα πρωτοβουλία πρέπει να συμφωνεί με το πρωτόκολλο 28 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα εγγυθούμε ότι δεν θα υπάρξει νέα πρωτοβουλία η οποία να έχει επιπτώσεις αναδρομικά για τους εταίρους και τους δικαιούχους. Σας ευχαριστούμε. Να μισή λεπτό κύριε Σομαγζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθε στην Επιτροπή των Περιφερειών έλεγα ότι ένας μικρός προπολογισμό για την Ευρώπη θα είναι πραγματικά μια τρομακτική έλλειψη φιλοδοξίας ε, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική και οι πολιτικές συνοχές δεν μπορούν να θυσιαστούν. Αν το κάνουμε αυτό, πραγματικά ε, δίνουμε τη νίκη στους ε, ευρωφοβικούς. Πρόκειται για ήττα. Αυτό θέλουν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Αυτά τα διδάγματα άντλησαν από τις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι το ερώτημα που του θέτω και λέω στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί περικοπές στον προπολογισμό της συνοχής, διότι περισσότερο από ποτέ τώρα θέλουμε περισσότερη συνοχή και οι περικοπές στον προπολογισμό της συνοχής θα σημάνουν λιγότερη εκπαίδευση για τους νέους, λιγότερη καινοτομία, λιγότερες επενδύσεις στις περιφέρειες λιγότερες θέσεις εργασίας και λιγότερη επιστηστική βοήθεια για τους ε, πιο ασθενείς ε, ενδέης. Ε, μεγαλύτερη διάσπαση και χάσμα μεταξύ των περιφερειών. Για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας είναι να ε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε έναν προϋπολογισμό επαρκή που θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στο βιωτικό επίπεδο ε, που πρέπει να φροντίσουμε και λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ κύριο Μαζέ. Κολάκουσιτς τώρα για ένα λεπτό. Αξιότιμε Πρόεδρε, εξωτιμοί ευρωβουλευτέ, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην ευημερία που να την προσφέρει εξίσου σε όλε τι χώρε μέλη. Αυτοί που έχουν αναπτυχθεί λιγότερο έχουν πολλέ οικονομικέ δραστηριότητε επειδή επεκτείνεται η αγορά. Αλλά εκεί που χώρε είναι λιγότερο αναπτυγμένε, όπω η Κροατία, δεν συμβαίνει αυτό. Και κυρίω στην ε, γεωργική παραγωγή η Κροατία Πέντε χρόνια τώρα από το 2013 έχασε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ κατά την ίδια περίοδο η Ρουμανία ε, πέτυχε συν 16 δισεκατομμύρια. Η κρατική δημοκρατία από τότε που έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισε 1,8 δις και στην Γεωργία έχασε 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι λογικό λοιπόν να ζητάμε οι πιο αναπτυγμένες χώρες να συνεισφέρουν περισσότερο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Κολακούσιτς. 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο. Σήμερα συζητούμε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία και επιβεβαιώνουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν και των ευρωεκλογών. Είδαμε ότι οι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν ε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, περιμένοντα περισσότερο. Οι αγρότες, οι επιχειρηματίε, περισσότερες στι πόλει, στην Ήπεθρο, περιμένουν περισσότερα, περισσότερε εξαγωγέ, καλύτερη έρευνα και καλύτερε. Ε, θέματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε καθήκον να τους ακούσουμε και να τους δώσουμε αποτελέσματα. Ο κόσμος περιμένει περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και το πρώτο μήνυμα προς, εμένα, προς εσάς κύριε Υπουργέ είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με πολύ λιγότερα. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι καινούριο πρέπει να διαθέσουμε κονδούλιο από κάτι που παίρνουμε. Δημιουργήσαμε το Ταμείο Επενδύσεων, το Connecting Europe Facility έχασε πράγματα. Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει οι νέε προτεραιότητε να χρηματοδοτούνται με νέου πόρου. Αλλιώ πρέπει να πούμε στου φοιτητέ ότι θα έχουμε λιγότερε υποτροφίε Εράσμου, στου γεωργού ότι οι ενισχύσει θα είναι λιγότερε και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δεύτερον, κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μου προ εσά είναι πότε θα είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είδαμε μέχρι τούδε από την Φιλανδική Προεδρία είναι ελάχιστα ψυχία και είναι πολύ λίγα. Χρειαζόμαστε τη δέσμευση σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του και πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε. Έχετε ευθύνη να μιλήσετε με το Κοινοβούλιο και αλλιώ πρέπει να το πω σαφέστατα. Το Κοινοβούλιο θα είναι υπεύθυνο και θα το κατηγορήσουν οι δικαιούχοι τη Ευρώπη αν δεν μπορέσουμε να του χρηματοδοτούμε μετά το 2021. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρισάν. Ένα λεπτό τώρα η κυρία Γκουαλμίνη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια γενική παρατήρηση και δύο πολύ σύντομα σχόλια. Καταρχάς το ψήφισμα είναι πολύ καλό. Συμμεριζόμαστε και εμείς την άποψη ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε με σθένους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένας θαραλέος προπολογισμό για την επόμενη επταετία. Πολύ καλή παράγραφος 5 που εισάγει μια αναθεώρηση των ίδιων πόρων ως στρατηγικό στόχο. Τώρα, τα δύο σχόλιά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέουμε σε οποιοδήποτε προπολογισμό και εσεί, κύριε Επίτροπε Χάν, το είπατε και μάλιστα με θετικό τρόπο στην ακρόαση. Ε, να υπάρχει σύγκληση μεταξύ των εσόδων και των εξόδων. Η πολιτική προπολογισμού δεν είναι μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία, δεν είναι μια μαθηματική απόδειξη, είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς αναθέτουμε πόρους προκειμένου να ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Είναι το επίκεντρο της δημοκρατίας μας και χωρίς αυτά οι δημοκρατίες μας δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Εάν λοιπόν η στόχη είναι φιλόδοξη η οικολογική μετάβαση, η εργασία των νέων, έρευνα, διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει να υπάρχουν και έσοδα τα οποία να είναι αυθεντικά ευρωπαϊκά. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μία αλλαγή νοοτροπίας, να κάνουμε ένα άλμα και να αλλάξουμε τα ευρωπαϊκά έσοδα. Δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε περισσότερους φόρους από του πολίτες. Ίσα ίσα θα μειωθεί η καθαρή συνεισφορά, αλλά να υπάρχει ένας εξευρωπαϊσμός των εσόδων, ένα ολοκληρωμένο όραμα των εισόδων και να μην είναι είναι πλέον ε, απλώς ε, ε, υπέρ των κυρίαρχων κρατών. Σας ευχαριστούμε πολύ για ένα λεπτό κύριο Στόρβαλτς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ του Πουράινεν, τι καλή συμβουλή μπορώ να δώσω στην Προεδρία αυτή. Τέσσερα πράγματα νομίζω. Πρώτα απ' όλα, Brexit. Χρειάζεται αλληλεγγύη και περισσότερα χρήματα από τις χώρες μέλη. Και πρέπει επίσης να σκεφτούμε την καινοτομία και την έρευνα. Εννοείται ότι πρέπει να τηρήσουμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για την έρευνα και την τεχνολογία. Δεύτερο, κι άλλοι το είπαν πριν από μένα, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε επενδύσεις. Επιγόντως μας χρειάζονται επενδύσεις. Υπάρχει μια πολύ ανησυχητική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, επενδύσεις και κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Χρειαζόμαστε δίκαιες λύσεις επίσης. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Οι οικονομικά, όσον αφορά την έρευνα, η πόρη διαφορετική. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ ακούς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστώ κύριο Άντρεσεν. Γιατί κάτι μου έμαθε, ότι το Συμβούλιο όταν δεν θέλει αυξήσεις είναι λαϊκιστικό. Εγώ ευχαρίστω να χαρακτηρίζομαι από εδώ και πέρα λαϊκιστή, γιατί πράγματι δεν θέλουμε δαπάνε υπερβολικέ από εδώ και πέρα. Αλλά τι είναι όμω, Δημαπο, γιατί είναι λαϊκισμό. Νούμερα ακούγονται συνεχώς σήμερα. Η Κομισιόν θέλει 1,1-1,4% του καθάριστου ε, εισοδήματος, το Κοινοβούλιο θέλει 1,3% ακούγονται ανώδυνα όλα αυτά. Μιλάμε για μικρά ποσοστά, μικρά νούμερα. Αλλά όμω κάνουμε του υπολογισμού, ε, τότε είναι 11 και 13%. Και αυτό πρέπει να πείτε στου πολίτε που θέλετε να απογραφείτε τι προσδοκίες τους, γιατί για τους πολίτες μιλάμε. Και αν μονίμως μιλάμε για αυξήσει και δεν το θέλει, σε καμία περίπτωση ο πολίτης, ε, τότε πραγματικά ε, στουρθοκαμιλίζουμε. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Όβεργκαρτ Νίλσεν. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι την εγκαταλείπει το Ενωμένο Βασίλειο που συνεισφέρει με πάρα πολλά χρήματα τα οποία θα λείψουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Η δημοκρατία μεταφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αύξηση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση των δαπανών που πάνε στην άμυνα, στο στρατό, τον ευρωπαϊκό, είναι πράγματα που δεν θέλουμε. Εδώ κάπου 20% θέλει αύξηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η αύξηση των μισθών μόλις και με έχει γίνει αισθητή τα τελευταία χρόνια. Είναι ντροπή και αγνοεί επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι με την αλαζονία παραβλέπουμε τον αγώνα των ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει να ε, πληρώνει για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ας αρχίσουμε να ξεφορτωνόμαστε τα 100, τις 130 λιμουζίνες που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και να επανέλθουμε σε φυσιολογικές πρακτικές που περιμένουμε και από οποιαδήποτε εταιρεία και επιχείρηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βαργκάρτ Νίλσεν, 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Χολμάιερ. Αξιότιμη Προεδρία του Συμβουλίου, αξιότιμη Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ, και ακούγοντα τι διάφορε προσδοκίε, νομίζω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ λογική. Τι θα πει λογική πρόταση. Έχουμε νέα καθήκοντα, άμυνα και αν άκουσα και τον προηγούμενο καλά κύριο ε, αυτοί δεν θέλουν φιλία και ειρήνη αλλά διαμάχηση για την παραθέση μεταξύ των μελών Θέλουμε λοιπόν ε, ένα λογικό προπολογισμό. Πρέπει να μιλήσω όμως για την έρευνα, τις επιστήμες, την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση. Ξέρουμε και είμαι υπερήφανη για την Βαβαρία, αλλά δεν ανατέλει πάνω από τη Βαβαρία μόνο. Ε, επομένως ε, πρέπει να έχουμε ουρανό και ήλιο σε όλη την Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη, ε, το Horizon 2020 είναι το κατάλληλο γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και πρέπει να συμφωνήσουμε. Επίσης έχουμε νομίζω κάποια καλύτερη κατανόηση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με τις προηγούμενες μεσομικές προοπτικές από Συμβουλίου, όχι όμως ό,τι αφορά τα κονδύλια. Αν έχουμε νέα και περισσότερα καθήκαντα, ε, τι θα γίνει. Ε, υπάρχει ανάγκη να ε, δοθούν και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι. Και νομίζω γι' αυτό και η θέση μας χαρακτηρίζεται στο Κοινοβούλιο από απόλυτη συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάιερ. Επόμενος, ο κύριος Λαρουτιγού, στο Δημοκράτης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, για να κερδίσουμε τη μάχη για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή μας λέει ότι κάθε χρόνο ότι λείπουν από 75 ε, έως 215 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα κερδίσουμε τη μάχη για το κλίμα αν δεν αυξηθεί ο προπολογισμό και αν δεν υπάρχει ένα κατάλληλο κλίμα το οποίο θα προστατεύει τους ε, μισθωτούς από την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση αν δεν έχουμε επενδύσει όπως πρέπει. Πρέπει να αυξηθούν από, από αρετήτως οι διπόροι. Το ο Ρούσβελτ είχε το κουράγιο το 1933 να αυξήσει τον προπολογισμό των ΗΠΑ και μάλιστα τριπλασίασε τον προπολογισμό με κατάλληλη φορολόγηση. Γιατί να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ε, οι φόροι για τα ωφέλη ήταν στο 45% και μειώθηκε στο 20% ενώ αυξάνουν τα μερίσματα. Γιατί να μην εφαρμόσουμε λοιπόν τις ιδέες του Ζακ Ντελόρ, του Μάριου Μόντι για ένα πραγματικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στους ιδίους πόρους και να έχουμε και ε, ομοσπονδιακό ε, καταμερισμό των εσόδων. Να έχουμε λοιπόν ένα πολύ πιο φιλόδοξο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριος Χόισικ από την ομάδα Renew. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο προπολογισμός θα είναι ουσιαστικός και θα είναι το καθημερινό μας ψωμί. Οι κίνδυνοι για όλη την Ευρώπη, για όλο τον πραλίτη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κλιματική κρίση, η α, καταστροφή της βιοπικιλότητας, η καταστροφή του Αμαζονίου και των δασών, οι τοξικές ουσίες, όλα αυτά είναι γύρω μας και αυτό όσο ο προπολογισμό είναι και μια ευκαιρία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, ε, καταστροφές και να τις αντιμετωπίσουμε ως ευκαιρία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για το κλίμα και τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να αποτελεί τη βάση αυτό και να είναι φιλόδοξε οι πολιτικέ μα, ώστε να ξέρει επίση και η δεξιά τι πει η αριστερά. Δεν μπορούμε να μιλάμε απλώ για το κλίμα και το περιβάλλον και μετά να τα καταστρέφουμε. Συνεχίζονται να γίνονται τέτοια πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε, μια βιομηχανία που δεν ρηπαίνει. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, τα ζώα, του γεωργού. Ο προπολογισμό αυτό δεν αφορά εμά. Το γεγονό ότι τα παιδιά μα πρέπει να έχουν ένα μέλλον και δεν μπορούμε να τα διαψεύσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Ακολουθεί ο κύριος Ντόρφμαν από το ΕΛΚΑ. Για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα είναι σαφές ε, ότι πρέπει ο προπολογισμό να βλέπει προς το μέλλον και να λάβει υπόψη τις προτεραιότητες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, έχουμε ε, την ανάγκη, είπατε εσείς, να κάνουμε κάποιες ε, περικοπές, να εξοικονομήσουμε και στη γεωργική πολιτική πρόταση. Μιλά για σημαντικές ε, εξοικονομήσεις στον τομέα αυτό και δεν τις δέχονται τις περικοπές τα κράτη-μέλη. Η πρόταση επίσης θα περικόψει πάρα πολύ και τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης. Το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αν λοιπόν κόψουμε πάνω από 40% τους πόρους αυτού του ταμείου, τελικά αυτά τα κράτη ε, τα οποία δεν θέλουν να πληρώσουν ε, τα πιο και τι θα κάνουν, θα βάλουν ε, για την εθνική του ε, γεωργική πολιτική ίδιους πόρους αυτά τα κράτη, τα φτωχότερα όμω κράτη δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν και αυτό δεν είναι δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Σαστέλα από το Ρινιού, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ψηφίζοντας σήμερα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες που να εκφράζει ότι οι προσδοκίες τους εισακούνται. Αλλά είναι και προειδοποίηση προς το Συμβούλιο, γιατί δείχνει την βούλησή μας να συμμετέχουμε πλήρως στη συζήτηση αυτή για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων μας στην ε, παραμονή ενός δύσκολου Brexit είναι κάτι που απαιτεί εξυγχρονισμό, απλοποίηση ε, των ιδιών πόρων αλλά και δημιουργία νέων ιδιών πόρων. Με ένα φιλόδοξο προπολογισμό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προτεραιότητε όσον αφορά το κλίμα, του νέου, την ε, κατάρτιση, την ενίσχυση τη Ευρωζώνης. Εξάλλου χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργητική πολιτική με φιλοδοξία για να προστατεύσουμε τους αγρότες μας και τα εισοδήματά τους προκειμένου να είναι σε θέση να παράγουν ασφαλή τρόφιμα σε καλές τιμέ και καλής ποιότητας που να σέβονται συγχρόνως και το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συνάλφα, Αντιπρόεδρε κάρα ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Όσκαρ Βάιλτ είχε πει ότι κοινικός είναι αυτός που ξέρει την τιμή όλων αλλά την αξία δεν τη γνωρίζει για τίποτα. Αυτό ταιριάζει στη σημερινή συζήτηση Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πούν ότι οι επενδύσεις ε, είναι δαπάνες, ε, είναι σπατάλοι και περιορίζουν ε, τις επενδύσεις που βοηθούν την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ασφάλεια, την άμυνα, την εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Δεν θέλω να τα αναγνωρίσουν, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τις προτεραιότητες. Θα ψηφίσουμε σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποιες ενδείξεις ε, ε, για το κατά πόσο θα ακολουθήσουμε το δρόμο της λογικής ή το δρόμο των αντικλήσεων παραθέσεων ε, και Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε όλη την ευθύνη για το μέλλον. δεν θα πρέπει να προδώσουμε το μέλλον μας. Τότε θα χαρακτηριστούμε προδότες. Πρέπει να προωθήσουμε την υπεραξία, την προσθέμενη αξία των δράσεών μας και εμείς είμαστε κύριε Επίτροπε στο πλευρό σας και θα σας στηρίξουμε στις ε, διαπραγματεύσεις που θα έχετε και εσείς να δώσετε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα στη δικασία ε, προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου από πλευρά χρόνου που τα πηγαίνουμε καλά, είναι σημαντική η συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη. Οπότε έχω την ε, δυνατότητα να δώσω το λόγο σε 7 συναδέλφου και θα ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο Μοντέρο Δε Αγγιλάρ, την κυρία Μοντέρο Δε Αγγιλάρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κοινή η αρμοδιότητα για τον καταρτήση του προπολογισμού ε, βάσει τη συνθήκη Λισαβόνας. Όσον αφορά τα όσα ψήφισε το Δεκέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επόμενο ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ ήταν απόλυτα σαφή. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση πολύ συγκεκριμένη ως απόδειξη και του σεβασμού και της αναγνώρισης ε, και του τομέα του τουρισμού. Ε, λυπάμαι που δεν είχαμε αυτή την πρόταση που διότι δεν την ήθελε ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη-μέλη. Ο διεθνής τουρισμός αυξήθηκε κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικός όχι μόνο για την Πορτογαλία αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος ε, ε, βοήθησε κάποιες χώρες να βγουν πιο γρήγορα από την οικονομική και επιστοτική κρίση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και ο τουρισμός, ο βιώσιμος τουρισμός να γίνει προτεραιότητα. Προχωρούμε με τον επόμενο ομιλητή από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι από τη Ρουμανία εγώ και νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε ε, τα σωστά ερωτήματα για να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε των πολιτών. Ο προπολογισμό αυτό πρέπει να καλύψει όσο γίνεται περισσότερε από τι ανάγκε των πολιτών, ώστε να μην πληρώνουν οι πιο αδύναμοι για του υπόλοιπου. Οπότε το ερώτημα είναι πώ κατανέμεται ο προπολογισμό αυτό. Θέλουμε περιφερειακά νοσοκομεία, θέλουμε αυτοκινητοδρόμους, θέλουμε καλό σύστημα υγείας, ε, γεωργία. Ωραία, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Ανάπτυξη, ε, γεωργία οικολογική, ε, έρευνα, καινοτομία κλπ. και Ναι, αλλά αν δεν ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες των πολιτών, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Οπότε οι διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, πρέπει να ξεκινήσουν. Μην ξεχνάτε ότι εδώ μα έχουν στείλει οι Ευρωπαίοι πολίτε και εγώ θα ψηφίσω ένα προπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε των συμπολιτών μου. Ευχαριστούμε τον κ. Τσιχοντάρου. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, πρέπει να σας πω ότι είναι πρόκληση να βρούμε ένα νέο επιτυχές οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη και τις χώρες μέλη που είναι εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι ένας απλός ε, τραπεζικός ε, προϋπολογισμός. Πρέπει να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες για ανάπτυξη των ε, εθνικών ΑΕΠ, αλλά να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των πολιτών, δηλαδή εκπαίδευση, ψηφιοποίηση, ασφάλεια και δεν πρέπει καν να υποτιμάμε την ε, πολιτική συνοχή και τη σημασία που έχει αυτή. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ την ιδέα που λέει ότι από 15 σε 35% ε, θα αυξήσουμε ε, τα προγράμματα. Εγώ πιστεύω στην συνοχή και στην αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Τόματσιτς. Από το ECR η επόμενη μιλήτρια. Σα ευχαριστώ. Η πρόταση για το πι έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στα μικρότερα, λιγότερα αναπτυγμένα κράτη-μέλη. Τα μηνύματα είναι ότι ουσιαστικά εγκαταλείπουμε τις προοπτικές ανάπτυξης για τα μικρότερα κράτη και δίνουμε μεγαλύτερη επιρροή στις μεγαλύτερες χώρες. Η πολιτική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να ενισχυθεί ιδίω σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση που στη χώρα από την Κροατία πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί πρόβλημα. Ε, μεταναστεύουν οι νέοι μας, οι μορφωμένοι νέοι μας φεύγουν από τη χώρα. Ε, πρέπει όμως να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη ζωή στην Ήπεθρο, να διατηρήσουμε υψηλά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θέλουμε μια ανταγωνιστική γεωργία. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το πετύχουμε αν δεν έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν είναι αποδεκτό λοιπόν και δεν θα πρέπει και κανένας να το δεχτεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Φερέρα τώρα από την ομάδα Γκου Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ασύμετρη ολοκλήρωση, δηλαδή τα ωφέλη και οι απώλειες των ευρωπαϊκών πολιτικών στο ενιαίο νόμισμα υποφελούν ε, τους ίδιους και βρίσκονται χαμένοι οι ίδιοι. Ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό πρέπει να προσπαθήσει να μειώσει τα χάσματα μεταξύ των χωρών μας, τις ασύμετρες επιπτώσεις της μετανάστευσης και να οδηγήσει σε πραγματικά ωφέλη. Λέει τα ίδια, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η συνοχή ποτέ δεν είχε τους κατάλληλους πόρους να κάνει τη δουλειά της. Ε, αντί να μειώσουμε λοιπόν το Ταμείο συνοχή. αυτό που κάνετε στην πραγματικότητα είναι ότι κάνετε περικοπές ε, για χώρες όπως η Πορτογαλία, για την οποία η πολιτική συνοχή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και φυσικά οι δικαιούχοι ε, θα είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες ε, προχωρούν τώρα προς ένα πιο στρατικοποιημένο ε, σύστημα, μία προσέγγιση που βλάπτει τη συνοχή. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να το απορρίψουμε. Δυστυχώς το ψήφισμα αυτό δεν είναι αρκετά ισχυρό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε, Ελκ Βάρμπο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πάντα μιλούσα υπέρ μιας αυστηρής ε, ε, πολιτικής ε, προϋπολογισμού, έναν ε, ε, στενό προϋπολογισμό. Το έλεγα πάντα ως βουλευτής στη χώρα μου και τώρα ως ευρωβουλευτής. Ήμασταν σαφείς στους ψηφοφόρους μας ότι δεν θα επιτρέψουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να διωγγωθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται και να δίνουμε και άλλα σουηδικά κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση επιτάπητος αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος κίνδυνος. Είναι 40% αύξηση της σουηδικής συμβολής στον προπολογισμό και είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα μπορούσα να δεχτώ. Ε, όντως είναι μεγάλε προκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ανταγωνιστικότητα κυρίω και δεν θα έπρεπε να πιέσουμε του πολίτε μα και του επιχειρηματίε μα να πληρώσουν ακόμα περισσότερου φόρου ώστε να χρηματοδοτούμε ε, την παραπάνω συμμετοχή στον ευρωπαϊκό κορβανά. Θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική μας, να επενδύουμε περισσότερο στην έρευνα, σε υποδομές ε, και στην αποτελεσματικότητα. Αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ε, ωφέλη και έτσι θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτε τη. Ευχαριστώ. Μάρκες ε, και είναι η τελευταία αυτή παρέμβαση από την ομάδα Σωστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, η Ευρώπη περνάει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της εξαιτία της ανεύθυνης κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι έτοιμη να τα χάσει όλα για εκλογικού λόγους και μόνο. Και θα το μετανιώσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν είναι σε θέση να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Η κίνδυνη είναι μεγάλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φτάνει προθεσμία και χρειαζόμαστε έναν ισχυρό προϋπολογισμό τώρα, ώστε να μπορέσουμε να ε, δώσουμε εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να πετύχουμε ανάπτυξη και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού όμως ακούμε ότι διάφορες χώρες στο Συμβούλιο θέλουν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στον προτινόμενο προπολογισμό. Όπως είπε και ο, πρόεδρο, ο, ο Επίτροπος και ο πρόεδρος Επιτροπής, τώρα πια έφτασε η ώρα. Πρέπει να στηρίξει το Συμβούλιο τις ίδιες θέσεις που στηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα ξέρουμε από πού έρχονται αυτές οι ιδέες για περικοπές. Εμεί χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με περισσότερη Ευρώπη και όχι με λιγότερο προπολογισμό, χαμηλότερο όπω προτείνουν διάφορε χώρε μέλη. Σας ευχαριστώ τη συνάδελφοι. Προχωρούμε με τον Επίτροπο Χάν. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσα πολύ προσεκτικά αγαπητοί ευρωβουλευτές τις παρεμβάσεις και δείχνουν ότι η τεράστια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προσιλωμένη στο στόχο ε, το ΠΔΠ να είναι φιλόδοξο, να εξασφαλίζει ένα βέβαιο μέλλον. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε με την επόμενη γενιά των προγραμμάτων. Αυτό θα είναι επιζήμιο, το χωροστάμε στους ε, πολίτες μας. Ε, να είναι προβλέψιμος ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η Ένωση θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ιδίως σε τομείς όπως είναι ψηφιακή κλιματική δράση, διαχείριση συνόρων και άμυνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φινλανδική Προεδρία για το έγγραφο που κατέθεσε χθε στην Κορεπέρ για την προετοιμασία της συζήτησης ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, για το επόμενο πιδελταπή. Καλό είναι που καταρτίστηκε αυτό το έγγραφο, αλλά για να το πω ξεκάθαρα, απογοητευτικά ήταν τα βασικά στοιχεία σε ό,τι το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού. Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί σε αυτή τη φάση των συζητήσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Καλούμε όμως την Προεδρία του Συμβουλίου και τους ηγέτες να λάβουν πλήρως υπόψη του στι θέσει του Ευρωκοινοβουλίου. Η Κομισιόν δεσμεύεται πλήρω να συνεργαστεί στενά με όλα τα θεσμικά όργανα και να διευκολύνει το διάλογο. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διαπραγματευτική του ομάδα ώστε οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ να ολοκληρωθούν έγκαιρα και μέσιο τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει εκ μέρους του Συμβουλίου κυρία Τουπουράινεν. Κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, εξότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολύ πολύτιμες απόψεις σας, τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις και τις σαφείς παρατηρήσεις σας. Πολλές από τις βασικές κοινέ μας προκλήσεις αναφέρθηκαν εδώ σήμερα στη συζήτηση και θα ήθελα απλώς να αναφέρω εδώ την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, τις επενδύσεις, ε, τη βιώσιμη γεωργία, τη συνοχή. Και τέλος, ε, κάτι εξίσου σημαντικό, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των κοινών μας αξιών. Είναι προφανές ότι αυτά είναι όλα προς το κοινό μας συμφέρον. Είναι τα πράγματα τα οποία απασχολούν τα θεσμικά μας όργανα, τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι οι κοινέ μας προκλήσεις. Και πρέπει να αντανακλώνται και στον κοινό μας προπολογισμό. Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να σέβεστε αυτές τις κοινέ προκλήσεις. Αλλά κυρίες και κύριοι, το ΠΔΠ δεν είναι απλώς μια λογιστική διαδικασία. Είναι ένα εργαλείο εφαρμογής και αυτό το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας αποφάσεις. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε και τι ε, συμβολή θα πρέπει να έχει το κάθε κράτος μέλος. Οι συνεισφορές των κρατών μελών πρέπει να είναι δίκες, πρέπει να είναι εφικτές και πρέπει να είναι και αποδεκτές από όλους, για όλα τα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω την σαφή δέσμευση της Φιλανδικής Προεδρίας ε, να συναντάτε τακτικά με την πραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Επιπλέον, ο τριμερίος διάλογος έχει ξεκινήσει σε πολλά τομεακά ζητήματα ήδη και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να ακούσουμε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτόν. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι εδώ σήμερα σε αυτή την Ολομέλεια συζητούμε το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο μαζί. Ανταλλάσσουμε απόψεις για το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θα προσαρμόσουμε λοιπόν το νέο πι χωρίς την κοινή μας προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμός μας είναι ο κατάλληλος για τη νέα περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και η δουλειά μας συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ και σας εύχομαι καλή επιτυχία τώρα στο πλαίσιο των συζητήσεων ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο της Μερσιάς Διάταξης. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της Μερσιάς Διάταξης, έκθεση της συναδέλφου Τούν σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του Ευρώ. Εδώ στο λόγο ε, στην κυρία Τούν για να μας παρουσιάσει την έκθεση της. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ένα νέο σύστημα με το οποίο μπορείτε να δηλώνετε την ε, το έτοιμά σας ε, για να λάβετε το λόγο στο πλαίσιο της δικασίας ε, ε, της μπλε κάρτας και της προσέξης προσοχής του Προέδρου και μπορείτε βέβαια και ηλεκτρονικά πατώντας το κουμπί με την κάρτα ψηφοφορίας από το μηχάνημα Γι' αυτό παρακαλώ να έχετε την, ψηφιακή, την κάρτα ψηφοφορίας μαζί σας. Αν δεν την έχετε μπορείτε με τον συνηθισμένο τρόπο είτε δηλαδή με το χαρτί, είτε αυτοπροσώπως εδώ να μας δηλώσετε. Θέλετε το λόγο. Και παρακαλώ να τηρούμε όλη το χρόνο αγόρευσης, γιατί έτσι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι θα μπορούν να πάρουν το λόγο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και τώρα προχωρούμε στην επόμενη συζήτηση. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιάννα Τούμ. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σας μιλήσω Να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ. Νομίζω αυτό είναι. Τώρα σα ακούω και εγώ καθαρά. Έλεγα λοιπόν ότι σα παρουσιάζω την έκθεση για την κοινωνική πολιτική στη ζώνη του Ευρώπου, που ε, έκρινε με μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή μας. Είμαι από την Εστονία και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργό μα είχε το προνόμιο μαζί με τον Ζακλόντ Γιούγκερ υπέγραψε τον πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ήδη από το 2017. Αυτό το φιλόδοξο έγγραφο που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει συγκεκριμένε αρχέ που πρέπει να τηρηθούν στι χώρε μέλη. Πρέπει να ευχαριστήσω την Επίτροπο Τάισεν για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει υπέρ των κοινωνικών πολιτικών παντού στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν εύκολο. Κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε τι κοινωνικέ προδιαγραφέ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος βγαίνει και λέει όχι. Και μετά έχουμε την αρχή της επικουρικότητας. Συγχρόνως όμως γνωρίζουμε ότι η κατάσταση κάθε άλλο παρά ιδανική είναι. Από το 2012 και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει αναχώρα συστάσεις όχι μόνο για τα οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά και για την κοινωνική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι μια διαδικασία χρήσιμη. Ε, Δυστυχώ το λέει και η έκθεση ότι το μέγεθος υλοποίηση των συστάσεων αυτών είναι πάρα πολύ χαμηλός. Υπάρχει κάποια μικρή πρόοδο μικρή, που αναφέρεται για το 72% των συστάσεων το 2012. Το 2018 το ποσοστό αυτό ε, κατέβηκε στο 39% χαμηλότερο από ποτέ. Οπότε ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μέτρα και να βρει τρόπο να πείσει τις χώρες μέλη ότι η κοινωνική υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου σημαντική όσο η εσωτερική αγορά ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, πρέπει επίσης οι συστάσεις αυτές να επεκταθούν και στις χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Χάρηκα που άκουσα ε, από την κυρία Φοντερ Λάιεν πριν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ομιλία που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποσχέθηκε ότι τις πρώτες 100 μέρες της θητείας της θα ε, προτείνει νέους νομοθετικούς μηχανισμούς έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν ελάχιστο εσόδημα. Και σε αυτούς που το σκέφτονται ακόμα και διστάζουν θέλω να πω ότι θα ληφθούν υπόψη εθνικές παραδόσεις και νομοθεσία που σημαίνει ότι κανένας δεν πρόκειται να παραβιάσει την αρχή της επικουρικότητας. Αλλά από την άλλη πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να βοηθηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και σε φτώχεια. Αλλιώ στην Ευρώπη θα καταλήξουμε να χάνουμε του ανθρώπου οι οποίοι θα φεύγουν να εργαστούν ε, αλλού και αυτό βέβαια δεν είναι προ όφελο ε, κανενό. Τώρα, στι ακροάσει του, διάφοροι υποψήφοι επίτροποι αναφέρθηκαν στον κοινωνικό πυλώνα και την επιθυμία του να λύσουν κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι με αναπηρίες, με χαμηλούς μισθούς, μειονότητες, κόσμος που ζει στη φτώχεια. Όλους αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και ακριβώς αυτό είναι που θέλουν οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και από εμά που τους εκπροσωπούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης για νέα προγράμματα κατά της ανεργίας που καλωσορίζουν τα συνδικάτα. Εμείς πήραμε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, για παράδειγμα, επιστολή που λέει ότι στηρίζουν την έκθεσή μας. Ε, αλλά συγχρόνως λέγανε πρέπει να στηρίξετε τη μία και την άλλη τροπολογία. Πάντως πιστεύω ότι πραγματικά κάνουμε κάτι καλό και βασίζομαι σε αυτήν την έκθεση και στη δικιά σας στήριξη σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφε και περνούμε στην Επίτροπο, την κυρία Τίσιν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται στο 7ο έτος σταθερούς ανάπτυξη, σταθερής ανάπτυξης και ε, όλο και περισσότεροι έχουν θέση εργασίας. Η φτώχεια μειώνει σε σταθερή ε, βάση, ε, βάση και καλών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένου οικονομικού στόχου και έχει καταφέρει να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οι κοινωνικέ και οικονομικέ ε, πολιτικέ είναι επίση όρει και μάλιστα προσφάτω έχουμε συμπεριλάβει και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ανάλυση και κοινή συνεννόηση σε στενό διάλογο με τα κράτη-μέλη και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, ωστόσο υπάρχουν ακόμα αποκλήσει ε, και μεταξύ χωρών αλλά και εντό των χωρών Υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες χώρες και σε άλλες ε, ε, παραμένει υψηλή ανεργία. Και η φτώχεια είναι ακόμα μια μεγάλη πρόκληση με έναν στους δέκα εργαζομένους να βρίσκονται στο ε, κίνδυνο φτώχειας. Εφαρμόζονται και νέες μορφές εργασίες οι οποίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και να στρεβλώσουν την αγορά. Επομένως, βασική μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι οι αγορές εργασίας να περιλαμβάνουν πολύ περισσότερους και να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι καλής ποιότητας. Περαιτέρω, οι γυναίκες εξακολουθούν να μειονεκτούν στην αγορά εργασίας παρά το γεγονό ότι υπάρχουν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στι γυναίκε από ό,τι στου άνδρε. Η μείωση αυτού του χάσματο θα ε, δημιουργήσει τεράστιε δυνατότητε και καλύτερε δυνατότητε για την οικονομία και για την κοινωνία. Θα υπάρχουν ε, ε δικαιότερε πολιτικέ ε, εξισορρόπηση οικογενειακού και εργασιακού βίου και λιγότερο αποκλεισμό προ αυτή την κατεύθυνση. Οι τεχνολογικέ αλλαγέ και η ψηφιοποίηση αλλάζουν επίση ει βάθο τη ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Είναι απόλυτα σαφέ ότι πρέπει πρέπει να αναβαθμίσουμε τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στις δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε τους ανθρώπους μας στις αλλαγές αυτές, σε αυτούς τους καιρούς και να μπορέσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, τις τεχνολογίες και επίσης να εξασφαλίσουμε και μια δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ε, ως προς το κλίμα. Το να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής μας είναι πιο επιτακτικό από ό,τι ποτέ. Μπορεί να μειώνεται μεν συνολικά η φτώχεια, ταυτόχρονα όμως ε, είμαστε μάρτυρας ε, μια πολύ, ενός πολύ μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων που εκφράζουν μια αίσθηση ότι είναι πιο ευάλωτοι. Υπάρχει ανισότητα, επισφάλεια στην αγορά εργασίας και αν, άνισος αντίκτυπος ε, της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών αλλαγών στις χώρες, στις περιφέρειες, στους τομεί και στους ανθρώπους οι επενδύσεις σε δεξιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν στις επόμενες κοινωνίες. Ε, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας επίσης θα πρέπει να ε, βοηθήσουν ε, και να προστατεύσουν τους πολιτισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Επιτροπή Απασχόλησης για αυτή την πολύ ισορροπημένη έκθεση η οποία παρουσιάζει πολύ καλά και τις θετικές αλλαγές αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και συμμερίζουμε τα βασικά συμπεράσματα. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια οικονομία κοινωνική αγορά που προστατεύει του πολίτε μα σε αυτού του καιρού αλλαγών και το να βοηθήσουμε στη σύγκληση, είναι ε, το κίνητρο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έχουν περάσει λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που ε, το προτείναμε και τώρα έχουν ξεκινήσει εφαρμογές και στις τελευταίες δύο διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι μισές ε, περίπου από τις συστάσεις αναχώρα, το 44% αφορούν προτεραιότητες του κοινωνικού πυλώνα. Έχουν προταθεί πολύ σημαντικά νομοθετικά μέτρα, κάποια έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνουν αρκετές αρχές του πυλώνα και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει για να μπορέσει μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πυλώνα και να υπάρχει συνδυασμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Ταμείων και κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επίση, ο πυλώνα βοήθησε στην αύξηση τη ποιότητα τη εργασία, σε επενδύσει και σε κοινωνική δικαιοσύνη και στι δίκαιε μεταβάσει στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου. Ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ένα από τα βασικά ε, κληροδοτήματα τη ε, αποχωρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πόρο απέχουμε έχουμε φυσικά από την ολοκλήρωση των εργασιών, όπω γνωρίζετε όλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πυλώνα ήρθε για να μείνει και να αποτελέσει επηξίδα για τι μελλοντικέ μα δράσει για την αποσχόληση και τον κοινωνικό τομέα. Επιπλέον, ξεκινώντα από το νέο κύκλο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα έχει νέα κατεύθυνση για να συμπεριλάβει και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ βάσει και τη συγκεκριμένη νομική βάση για τα θέματα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες ώστε να έχουμε μια κοινωνία που περιλαμβάνει πολύ περισσότερους και να είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει τις αλλαγές. Οι ισχυρότερες κοινωνίες θα ενισχύσουν φυσικά και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Ευρωζώνη και θα ανοίξουν το δρόμο για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Όπως ξέρετε, η εφαρμογή των αρχών του πυλώνα επιτόπου, καθώς επίσης και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μια κοινή απόπειρα, την οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μείνει στην πρώτη γραμμή για να προωθήσει τη σύγκληση των κοινωνικών ε, συνθήκων και των συνθήκων διαβίωσης σε όλη την Ευρώπη και θα υποστηρίξει τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις ε, και τις περιφέρειες σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπη. Στην συζήτηση τώρα τη γενική, τον λόγο πρώτη θα λάβει η κυρία Μαρία Γουόλς από το ΕΛΚΑ. Ένα μισή λεπτό. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω την Γιάννα Τούμα και τους άλλους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και ιδίω συναδέλφου μου από το ΕΛΚΑ. Επίση, πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνικέ και οικονομικέ πολιτικέ να λειτουργούν παντού και να μην είναι αντιφατικέ μεταξύ του, να πηγαίνουν δηλαδή προ την ίδια κατεύθυνση. Η έκθεση αυτή συνεχίζει να δίνει προσοχή σε κάποια επίμονα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ε, μειώσουμε την ανεργία των νέων, να, ε, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια ιδίω των παιδιών, να έχουμε ισότιμη συμμετοχή στην αγορά, ισότητα όλων των μελών τη κοινωνία, να προωθήσουμε επίση την ανταγωνιστικότητα αλλά και να σκεφτούμε το μέλλον και πώ θα προσαρμόσουμε τι δεξιότητε και τα κοινωνικά συστήματα και μιλώ ιδίω για τι αστικέ και τι αγροτικέ περιοχές. Πρέπει αυτά όλα να είναι προτεραιότητε τα επόμενα χρόνια. 10 Οκτωβρίου είναι η μέρα ε, για την ε, ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ψυχική υγεία. Είναι λυπηρό που η Ένωση εστιάζει πολύ λιγότερο τα πρόσφατα χρόνια στην ψυχική υγεία. Παρά το κόστος και το ατομικό και το οικονομικό το γενικότερο, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί κονκίνων και πολύ και στον τομέα αυτό. Δεν θα φροντίσουμε την υγεία των πολιτών αν δεν φροντίσουμε, αν δεν ασχοληθούμε με την ψυχική υγεία. Τα κράτη-μέλη πρέπει όλα να μπορούν να βελτιώσουν τις πολιτικές ψυχικής υγείας και ζητούμε εδώ στην έκθεση συγκεκριμένα μέτρα πρόωθηση, ε, μέτρων και προληπτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ε, η υγεία και η θέση απασχόλησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Θέλω να ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την Γιάννα Τούμ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γουόλς. Ναι, να υπάρξει και ο χρόνος για τα χειροκροτήματα. Και να δώσω τώρα στην κυρία Γιονγκέριους, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ένα πλονόμισμα ή μία αγορά. Πρέπει να έχει και μια άλλη διάσταση για το μέλλον. Και γνωρίζουμε για τις νέες τεχνολογίες, για την οικονομική ανάπτυξη για την δίκαια μετάβαση που απαιτείται εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Και αυτά πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσουν. Δεν μπορεί να ε, διχαζόμαστε. Όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ε, τομείς. Όλοι. Και ο καθένας μπορεί κάτι να προσφέρει. Είναι μια καλά ισορροπημένη η έκθεση αυτή που θα ψηφίσουμε σήμερα. Γιατί ακριβώς αυτό προσπαθεί να πετύχει. Η Ευρώπη των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πρέπει να προσφέρει καλύτερη κοινωνική προστασία. Και πρέπει γρήγορα να τελειώσει αυτή η αδικία του χάσματος στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους ε, ανθρώπους που είναι μεγαλύτερη ηλικία και να προσφέρουμε περισσότερες προοπτικές για εργασία στους ε, ανάπηρους και στους πιο αδύναμους για να μπορέσουν και αυτοί να ανθίσουν στο χώρο εργασίας. Χρειάζεται κατάλληλη κατάρτιση επίσης για να μπορούν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το μέλλον με εμπιστοσύνη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε κάποιες ιδέες για την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω όντω να προχωρήσει. Αλλά θα πρέπει και οι χώρε μέλη να συμφωνήσουν, το Συμβούλιο. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και μόνο τότε θα αντιμετωπίσουμε τη μακροχρόνια ενέργεια και μόνο τότε θα στηρίξουμε τι πιο ευάλωτε περιφέρειε. Τότε μόνο θα μπορεί να πει ο καθένα στην Ευρώπη ότι η Ευρώπη είναι και δικιά του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιγκέριος. Επόμενη Σιλβί Μπρινέ για την ομάδα Renew Europe. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τούμ για την εξαιρετική της έκθεση και χαίρομαι που το Ευρωκοινοβούλιο στην πλειοψηφία του είναι υπέρ της έκθεσης αυτής ε, για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ε, Ευρωζώνης. Έκθεση που έχετε σε συνέχεια των ειδικών στάσεων αναχώρα που δημοσίευσε η Κομισιόν τον Ιούνιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι γενικοί προσανατολισμοί τη έκθεση δείχνουν ότι ε, το νέο κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, με έμφαση στις επενδύσεις. Θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία. Πρώτον, το αίτημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την κατάθεση ενός νομικού μέσου ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση να έχουν ένα κατώτατο δίκαιο μισθό με σεβασμό στι εθνικέ παραδόσει. Αυτό είναι κάτι μείζωνο σημασία. Εγγράφεται στου πολιτικού προσανατολισμού τη Ούρσουλα Φοντρελά ενό προτεραιότητα για την επόμενη ε, κοινοβουλευτική περίοδο σε διαβάτη κοινωνική συνοχή. Και είναι, κατά την άποψή μου, και μια απάντηση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλά κράτη-μέλη. Το δεύτερο σχολείο μου έχει να κάνει με του εργαζόμενου σε πλατφόρμε και τι συνθήκε εργασία του γνωρίζουμε ότι η εργασία που γίνεται μέσω αυτών των διαδικτυακών πλατφορμών που είναι καλό έχει αυξηθεί κατά 25% και παραπάνω τα τελευταία χρόνια και αφορά πλέον περίπου 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ενώ υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που μεμονωμένα έχουν εφαρμόσει εθνικά μέτρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ε, το στίγμα και την κατεύθυνση που θα εξασφαλίσει την κοινωνική προστασία αυτών των εργαζομένων. Εγγυόμενοι όλα τους τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπρίνη. Προχωρούμε εκ μέρους των Πρασίνων και της Ελεύθερης Επικής Συμμαχίας ε, Πέτερ Χάνσεν για 1,5 λεπτό. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει σε αυτό το φάκελο. Εμεί οι πράσινοι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την έκθεση και κυρίω επειδή καλύπτει διάφορα κοινωνικά ζητήματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν στην επόμενη θητεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η έκθεση στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινωνικού στόχου, κοινωνικέ προτεραιότητε ε, στο νέο πλαίσιο και επίσης όσον αφορά τους ε, πόρους, τους κοινωνικούς που θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο προπολογισμό. Από πλευρά των πρασίνων είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και η αδικία που υπάρχει μεταξύ των ε, γενεών. Λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως ε, θέλουμε να προχωρήσει και η διαφάνεια να μην υπάρχει πια αυτό το χάσμα στις αμοιβέ μεταξύ αντρών και γυναικών. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις συντάξεις, έτσι. Ε, χαιρόμαστε που η έκθεση αυτή ζητάει λύσεις για να αντιμετωπιστεί μακροχρόνια ανεργία, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και επίσης ζητάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διασφαλιστούν και οι εργαζόμενες στις πλατφόρμες, ανεξάρτητα από το καθεστώς εργασίας που έχουν. Θα παρακολουθούμε λοιπόν την Επιτροπή και το νομοθετικό της έργο και τις νομοθετικές της προτάσεις τα επόμενα χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε και δεν το λόγο στην κυρία Φαζαμέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Συγήτρια, όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει καλύτερα. Και κύριε Συγκίντρια, δεν έχετε δίκιο. Αντίθετα, αποτελείται από οικονομίε εντελώ διαφορετικέ μεταξύ του, με κοινωνική και οικονομική και ρυθμιστική κατάσταση τελείω διαφορετική τη μια από την άλλη. Η έκθεσή σα είναι γεμάτη ιδεολογία και μεροληπτή. Ε, περιλαμβάνεται και την Τουρκία στα δεδομένα σας και αυτό ε, συνεχώς με την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας σε βάρος των ε, πιο αδύναμων συμπατριωτών μας. Συνεπώ, φυσικά και θα καταψηφίσουμε την έκθεση αυτή και θα στηρίξουμε τον αλλακτικό ψήφισμα του συναδέλφου Τζιντοράιλ, γιατί είναι πολύ πιο αναγκαίο να έχουν την κυριαρχία του οι χώρε μέλη όταν πρόκειται για την οικονομική και κοινωνική πολιτική και επειδή πρέπει να μπορούν να θέσουν τις προτερότητε τους βάζοντας τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται για την απασχόληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ECR, κυρία Ζαλεύσκα, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς βεβαίως και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την εντατική δουλειά για την ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής που είναι κάτι ενδιαφέρον σίγουρα για την ζώνη του ευρώ. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η φτώχεια, κοινωνική ανάπτυξη, οι ε, νέοι. Ε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ακολουθήσει η κοινωνία την επανάσταση του 21ου αιώνα. Φαίνεται να υπάρχουν λίγες ιδέες ε, για το πώς ε, μπορεί να προσαρμοστεί η κοινωνία μας, ε, να εκπαιδευτούν οι νέοι μας και όλοι οι πολίτες. Και δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει ιδέες προς αυτό. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη παρέμβαση στην ένωμη τάξη από την Ευρώπη Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε ειλικρινά για λύσεις και όχι να περιγράφουμε απλά την κατάσταση. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Γκουέντζιέλ, η κυρία Περέρα, 1,5 λεπτό. Καλημέρα. Η κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές ε, οι οποίες επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται βάσει μια συνθήκη η οποία τελικά ποινικοποιεί οποιαδήποτε αριστερή ή προοδευτική πολιτική. Από τότε που ενταχθήκαμε στο ευρώ, αυτό σημαίνει ότι όπω θα δρομούμε κοινωνικά, έχουν ε, μείνει στάσιμοι οι μισθοί, υπάρχουν προβλήματα με την εργατική τάξη, υπάρχουν προβλήματα με την ένταξη των μεταναστών. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μπορούμε να δεχτούμε το πιο αυστηρό ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά οικονομικά. Η χώρα μου στο παρελθόν τα δέχτηκε όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ταυτόχρονα να αυξάνουμε ε, τις φόρους, ε, να έχουμε χειρότερες ε, δημόσιες υπηρεσίες και να μην υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ε, και δεν μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους γυρεότερους σεβόμενοι και τους αυστηρούς πολιτικές του ευρώ αυτοί που βρίσκονται στη δεινότερη θέση και έχουν τη λιγότερη οικονομική ευχέρεια θα βρεθούν στη δεινότερη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Τσεχόφσκι έχει ε, μπλε κάρτα για σας. Τη δέχεστε? Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Σντεχόφσκι. Από το όνομα του ΕΛΚ. Όχι. Να προχωρήσουμε με την κυρία Γκέμα από τους μη γεγραμμένους. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Οι πολιτικές στήριξη του ισοδύναματος σε πολλές χώρες όπως και η Ιταλία ήδη βοηθάει τους ε, πιο ευάλωτους ε, του πληθυσμού. Αλλά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις παρεφές τους ε, φτώχειας και οι οικονομικές ανισότητες αυξάνονται συνεχώς. Η οικονομική κρίση έπληξε περισσότερους αυτούς που είχαν ήδη δυσκολίες και εδώ θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχει αναλάβει δράση και ανέπτυξε την ε, μεγάλη της ανησυχία την ε, σαρνιτικής ε, συνέπειες που έχουμε λόγω της λιτότητας και επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να τους εγγυηθούμε μεγαλύτερη ποιότητα ζωής. Η δέσμευσή μου θα είναι συνεχής και θα είναι πάντα προς την κατεύθυνση ενός σχεδίου κοινωνικής προστασίας που θα εγγυάται απολύτως ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής και κυρίως θα σέβεται το δικαίωμα των ατόμων αυτών στη διαφορετικότητα και όχι στην ισότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προχωρούμε με τον συνάδελφο Ράτκη από την ομάδα του ΕΛΚΑ. Ένα λεπτό. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω θέρμα καταρχάς την εισηγήτρια για τη δουλειά της ε, που ήδη από την αρχή της ε, θητείας αυτής ε, λέμε ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλο στένος την επόμενη πενταετία για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια ο Πρόεδρος Γιουνκέρα. Θέλω να το πω ξεκάθαρο ότι στην ομάδα μας σε ό,τι αφορά το σύστημα αντασφάλισης ανεργίας, ε, τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Η γερμανική αντιπροσωπεία ε, το βλέπει με κριτικό πνεύμα ε, και πρέπει να σας πω ότι θα το μελετήσουμε και παρόλα αυτά με κριτικό πνεύμα εξακολουθούμε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το θέμα. Σίγουρα παρόλα αυτά πρέπει να στηριχτεί η απασχόληση των νέων, να καταπολεμηθεί η νεανική ανεργία, πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει και μεγάλη φτώχεια και είναι κάτι που για το ΕΛΚΑ ε, είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, να κάνουμε βήματα, αλλά βήματα προς αυτά τα οποία η ομάδα μας θεωρεί ότι είναι προς την που η ομάδα μας θεωρεί να είναι σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκουαλμίνη τώρα, σοσιαλιστές και δημοκράτες. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή και πολύ αποτελεσματική και φέρνει στην επιφάνεια τα ανησυχητικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Χώρου Εργασίας αλλά ταυτόχρονα αναφέρει και το στόχο του 75% ως ποσοστό μέσης απασχόλησης. Εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι γιατί αμφισβητούμε καινοτόμα και ουσιαστικά μέτρα όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ένταξης ε, ε, για να καταπολεμήσουμε την ανεργία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ε, το οποίο άλλωστε η Ούρσουλα Φαντερλάιν έχει συμπεριλάβει στις 100 μέρες της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς να αμφισβητούνται οι πόροι και το αίτημα για ένα χρηματοδοτικό μέσο για τα εξωτερικά σοκ και τις επιχειρηματικές κρίσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, Ευρώπη της εργασίας, μια κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στη στρατηγική του Άμστερνταμ, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση του 1997 ε, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο μια οικονομική Ευρώπη, πρέπει να είναι μια κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη τη εργασία. Σα ευχαριστώ. Προχωρούμε με την συνάδελφο Λάγκεν Ζήπεν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας ημέρα. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις που έρχονται στην κατάλληλη στιγμή, τοπίζουν τα σωστά προβλήματα και ζητούν τη σωστή αντιμετώπιση. Μία από τις εκθέσεις αυτές είναι η εκθέση της κυρίας Τούμ και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τούμ. Εδώ θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και δεν το λέω μόνο γιατί είμαι και εγώ προσωπικά ένα από αυτά τα άτομα, αλλά γιατί εδώ μιλάμε για την απασχόληση και πράγματι για τα άτομα με αναπηρία η έκθεση εκφράζει τη λύπη για το ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η πρόσβαση, η ένταξη είναι ανθρώπινα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και έχουμε και ε, επικυρώσει την Σύμβαση 2010 και η μη κριτική μεταχείριση είναι προτεραιότητα. Το αναφέρει αυτό, το τονίζει η έκθεση η οικονομική και κοινωνική πολιτική στην Ένωση θα πρέπει να συμβαδίζουν χέρι-χέρι. Ο κοινωνικό προπολογισμό πρέπει να είναι επαρκή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ράιλ από την ομάδα ΙΝΤΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρώπη σίγουρα είναι πολύχρωμη, είναι πολυεπίπεδη, πολύμορφη και αυτό πρέπει να διατηρηθεί γιατί είναι η ισχύ μα. Ο προγραμματισμό, ο σχεδιασμό, η συγκέντρωση δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε κατά του συστήματο αντασφάλιση ανεργία γιατί υπάρχουν τελείω διαφορετικέ παραδόσει και καταστάσει, άρα χρειάζονται περιφερειακέ λύσει. Επίση αρνούμαστε και τον κατώ μισθό. Θέλουμε ένα γερμανικό, αλλά όχι ευρωπαϊκό, γιατί αυτό θα δημιουργήσει στρεβλώσεις. Επίσης, ευρωπαϊκή εγγύηση για την των παιδιών. Φυσικά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αλλά ήδη υπάρχουν τρία ταμεία τα οποία δεν έχουν φέρει τίποτα. Και εγώ ως παιδί ε, αντιμετώπισα την ε, φτώχεια και πάρα πολλά παιδιά στην ε, χώρα μου και μας βοηθούσαν οι ενόριστοι τα λοιπά. Δεν λύνονται τα προβλήματα όμως με τον τρόπο αυτό. δεν μπορούμε να το λύσουμε δίνοντας κίνητρα στους στοχούς που κάνουν συνέχεια παιδιά η κοινωνική πολιτική δεν είναι αυτή που θα ε, μοιράζει λεφτά ε, σε όσους δεν δουλεύουν, αλλά σε αυτούς που δουλεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Ραφάλ Σκαϊσιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πολιτική στρατηγική ε, στο κοινωνικό τομέα σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα έχουμε πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές είναι το δημογραφικό, γύρανση του πληθυσμού, είναι η ψηφιοποίηση, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η Ευρώπη το αρνείται αυτό εδώ και 10 ε, χρόνια. Ο αριθμός του πληθυσμού που είναι πάνω από 65 αυξάνει συνεχώς σε όλες τις χώρες. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα ε, καλύτερης προσφοράς ε, υπηρεσιών υγείας αλλά και πολύ χαμηλού αριθμού γεννήσεων. Η Ευρώπη λοιπόν ε, πρέπει να αντιμετωπίσει την ε, περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων. Χρειάζεται μια καλύτερη στρατηγική για την πρόσβαση επίσης μακροπρόθεσμα στα συστήματα υγείας. Ε, πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις μικροεπενδύσεις, αλλά και την αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχουν καλές προδιαγραφές ε, για τους εργαζόμενους και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την συνεργασία σας μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Έτενταλ, ε, όχι, συγγνώμη, διορθώνω. η κυρία Ροντινέλη έχει το λόγο, κυρία Σπίτενταλ που είπα, είναι μετά. Ροντινέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την έκθεση που λέει τα πάντα και είναι και αντίθετο με τα πάντα. Αντί να υπάρχουν επενδύσεις για την ε, κοινωνική πολιτική, για την απασχόληση και την κατάρτιση και σας διαβάζω εδώ την παράγραφο 2, ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει απαραίτητο στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις συστάσεις αναχώρα, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτές τις πολιτικές λιτότητες οι οποίες περικόπτουν το, κράτος, ε, το κοινωνικό κράτος ε, και την ένταξη των τελευταίων και των λιγότερο ευνοημένων. Αυτή είναι μια τεράστια πολιτική αντίφαση η οποία δεν είναι πλέον αποδεκτή στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεν αρκεί να μιλάμε για κατώτατο μισθό και για απασχόληση των νέων όταν μετά δεν υπάρχουν επενδύσει για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Υποβάλαμε στην Επιτροπή Τροπολογίε, πολλέ από τι οποίε έγιναν αποδεκτέ, αλλά δυστυχώ δεν αρκούν για να αλλάξουμε αυτό το φιλελευθερικό και αυστηρό πλαίσιο που μας ζήτησαν οι πολίτες μας να διακόψουμε υπέρ της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της ισότητας για όλους. Το κίνημα Πέντε Αστέρια λοιπόν θα πόσχει από αυτή την έκθεση η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ροντινέλη. Τώρα η κυρία Σχετένταλ εκ μέρου του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. πολύ ασχοληθήκαμε με τα νομικά ζητήματα ε, που γύρονται με αυτή την κοινωνική πολιτική. Φορολογούμενοι θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν ε, για άλλους ε, υπηκόους άλλων κρατών. Τώρα όμως με τον κύριο Τίμερμανς ε, στην κορυφή. Βλέπουμε ότι θέλει αυτή την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση. Ουσιαστικά αυτό θέλει να πετύχει με το σύστημα αντασφάλισης ε, για την ανεργία. Εμείς πάντοτε ήμασταν αντίθετοι σε κάτι τέτοιο και θεωρούμε ότι τα νέα ε, νομοθετήματα ουσιαστικά μας γυρίζουν σε σοσιαλδημοκρατικές ε, φιλοδοξίες. Να πληρώσουμε όλοι ε, για τα κοινωνικά ελλείμματα ορισμένων χωρών. Δεν θα πρέπει να καταβάλουν χρήματα αυτοί που πληρώνουν για τα ταμεία της δικής τους ασφάλισης και να βάλουν το χέρι στη τσέπη για άλλες χώρες. Άγιου Σαλίμπα από την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει ότι οι οικονομικέ συνθήκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευνοϊκέ και ότι τα ποσοστά απασχόλησης ανεβαίνουν συνεχώς. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά τον πλούτο και διαφορές στα εισοδήματα, κάτι το οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων. Η φτώχεια μέσα στην εργασία, η επίτευξη ε, αξιοπρεπών συνθήκων ζωή, η ποιότητα τη εργασία, καλή μισθή, είναι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Δεν φτάνει να έχει κανεί μια δουλειά πρέπει να έχει και μια αξιοπρεπή ζωή συγχρόνω με τους φίλους του και τις οικογένειές του. Χρειαζόμαστε λοιπόν εργασιακές πολιτικές που να βελτιώνουν τις ηθίκες εργασίας και να προσφέρουν δίκαια απασχόληση και απασχόληση ποιότητας για όλους τους Ευρωπαίους. Για πρώτη φορά με την έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα υιοθετήσει την ε, ιδέα του δικαιώματος να μπορεί κανείς να αποσυνδεθεί ψηφιακά είναι ένα πρώτο βήμα ε, για το δικαίωμα αυτό, για να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στον ιδιωτικό βίο και την εργασία. Όταν ε, συζήτησα γι' αυτό για πρώτη φορά ήταν ένα ταμπού το να μπορεί κανείς να αποσυνδέεται μετά την δουλειά του. Αλλά τώρα θα γίνει σύσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση θέλω να πω ότι στηρίζω και την αντασφάλιση ανεργία σαν ένα νέο μέσο για να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανεργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε με την κυρία Ντούρη Νικολ, Νικολσόνοβα. Ένα λεπτό. ECR. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για την επιτυχία στην απασχόληση και να κοιτάξουμε τις συνασχετικές μελέτες που λένε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της γύρανσης του πληθυσμού, ούτε του κλίματος, ούτε των ψηφιακών αλλαγών. Το κόστος των αλλαγών αυτών θα μας έρθει και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο αυξάνοντα ε, τα κονδύλια. Σύμφωνα με τον ε, όσα 70% της απασχόλησης ε, στην Ευρώπη κινδυνεύει από τον αυτοματισμό. Η απειλή αυτή είναι πολύ μεγάλη, 10% στην Φιλανδία αλλά 30% ε, στην χώρα μου την Σλοβακία. Το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού δεν έχει καθόλου προσόντα ε, ψηφιακά και η μετάβαση αυτή βέβαια θα επιβαρύνει κυρίως τους πιο αδύναμους στις κοινωνίες μας. Τι χρειάζεται λοιπόν, καινοτομία, παραγωγικότητα, κοινωνικά δικαιώματα, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η κοινωνική Ευρώπη θα ανθίσει μόνο εάν οι οικονομικέ μας πολιτικέ δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον. Έχουμε τον ίδιο στόχο, οπότε ας σταματήσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στην ιδεολογία ή σε πολιτικά πυροτεχνήματα, αλλά ας φροντίσουμε όλοι μαζί για τη σωστή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και ο Στεχόσκι από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε να σας ευχαριστήσω να ευχαριστήσω όμως πρώτα απ' όλα τη Γιάννα Τούμ για την έκθεση αυτή. Είναι μια έκθεση ποιοτική κατά την άποψή μου, αλλά υπάρχει ένα θέμα που θέλω να θέσω. Στο ένα, η Γιάννα Τούμ λέει ότι θέλει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την αντιμετώπιση μακροχρόνιας ανεργίας. Μα έχουμε το αναθεωρημένο έκτα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ρωτώ λοιπόν, από πού θα βρούμε χρήματα για αυτό το νέο μέσο που θέλετε να θεσπιστεί. Έχουμε ήδη δύο εργαλεία, τα οποία λειτουργούν καλά και θα τα αποδυναμώσουμε βάζοντας χρήματα σε κάτι καινούριο, σε κάτι πρόσθετο. Δηλαδή αντί να την απλουστεύουμε, την κάνουμε πιο πολύπλοκη την Ευρώπη τελικά δημιουργώντας κάτι που ουσιαστικά έρχεται σε ανταγωνισμό με κάτι που ήδη φύσταται. Δεν νομίζω ότι αυτό δίνει την απάντηση στο πρόβλημα αυτό, γι' αυτό και δεν μπορώ να στηρίξω το συγκεκριμένο κομμάτι της έκθεσης, αν και την έκθεση θα την υποστηρίξω. Πρόεδρο σας, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινούμε ε, στο Κατσδιάι με τον συνάδελφο Κάνεφ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στηρίζω την ε, έκθεση αυτή παρόλο που περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία. Πιστεύω ότι οι προτάσεις αυτές, οι τόσο αντιφατικές, θα πρέπει να συζητηθούν εδώ στο σώμα και σίγουρα ε, θα υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ των ε, χωρών, μεταξύ των πολιτικών ομάδων που έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Όμως, η έκθεση υπογραμμίζει πάρα πολύ την περίπτωση των πιο αδύναμων, των πιο ευάλωτων ανθρώπων ή ε, μιλάει πολύ για τις χώρες ε, που έχουν περισσότερα προβλήματα και αδυναμίες. Δεν πρέπει όμως συγχρόνως να ξεχνάμε και τα προβλήματα στην αγορά εργασίας. Είμαι από την Βουλγαρία, όπου τα έσοδα είναι πιο χαμηλά και όπου οι πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού είναι πολύ άριθμες. Ελπίζω οι προτάσεις να προχωρήσουν και να αρχίσουν να ισχύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι κοινωνικέ ε, πολιτικέ πρέπει να εφαρμόζονται επίση όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η Επιτροπή. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Στον προπολογισμό αυξάνεται τις δαπάνες της ε, άμυνας από 15 στα 30 εκατομμύρια. Γιατί αυτά τα χρήματα να μην πάνε στην καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Γιατί τα χρήματα αυτά πηγαίνουν ε, σαν ενίσχυση ε, του στρατού. Γιατί δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε ασφάλεια αλλά εκτό από την ασφάλεια, χρειαζόμαστε και αξιοπρεπή ζωή. Χρειαζόμαστε ασφάλεια για να μπορεί κανεί να ζήσει, για να μπορεί να αγοράζει ε, φαγητό. Αυτό είναι ασφάλεια. Η εξασφάλιση αυτών των αναγών. Προστασία από την τρομοκρατία, ναι, αλλά μήπω να ελέγξουμε καλύτερα τι εξαγωγέ όπλων από την Ευρώπη, για να μην βοηθάμε ε, μερικέ χώρε να βομβαρδίζουν άλλε. Έτσι θα φέρουμε την ειρήνη και όχι στηρίζοντας οικονομικά την αμυντική βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε να πάρουμε ε, όσο το περισσότερο χρόνο για να δώσουμε το λόγο στη στο πλαίσιο τη δεκαετία προσέγγιση Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε ενδιάμεσε ε, ερωτήσεις κύριε Στεχόφσκι. Επόμενη από τις σοσιαλιστέ και Δημοκράτες κυρία Γουόρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την επόμενη πενταετία το Ευρωπαϊκό όραμα πρέπει να στηθεί σε μια προοδευτική πλατφόρμα η οποία θα περιλαμβάνει και οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Χωρίς μια τέτοια πλατφόρμα θα συνεχίσουν να υπάρχουν διακρίσεις και ανισότητες στο εργατικό δυναμικό αλλά και στους μισθούς. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τις εισοδηματικέ ανισότητες και να υπάρχει αύξηση εισοδημάτων για τα μεσαία και τα κατώτερα στρέμματα και να υπάρχουν και ε, κατάλληλη προετοιμασία για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και να μην υπάρχουν και κενά στα συντοξιοδοτικά. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δεμάτων είναι δικό μα πυλώνα εδώ στι Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε και υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία να έχουμε το πρώτο ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να μπορεί να λαμβάνει κάποιο αρκετά ώστε να μπορεί να επιβιώνει. Για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επενδύσουμε στου ανθρώπου. Και τα δύο είναι αλληλένδετα και αν δεν μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αδικίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τόματσιτς, ένα λεπτό. Ε, ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κροατική κυβέρνηση έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Εγώ δεν τα σημερώζω με αυτά τα σχέδια, δεν πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Η Κροατία απέχει πάρα πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αντιμετωπίζουμε και μία νέα ύφεση η οποία είναι πρώτων πυλών. Πολλές περιοχές της Ευρώπης ακόμα έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ ε, μεγάλη μακροχρόνια ανεργία και μετανάστευση. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κροατίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μετατοπίσουμε τη φορολόγηση σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές ε, και να υπάρξουν ε, νέες ε, ε, φορολογικές πολιτικές ε, ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει να δίνονται στα κατάλληλα μέρη. Θα πρέπει να υπάρχει αξιοπρεπής τρόπος διαβίωσης για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Επόμενος, επόμενη κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφερόμαστε ε, στις κοινωνικές πολιτικές και την απασχόληση στην Ευρωζώνη και θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ιρλανδία. Προσπαθούν με να παρουσιάσουν την ε, απασχόληση στην Ιρλανδία με αισιόδοξο πνεύμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά συμβόλαια μηδενικών ορών, επισφαλής ε, θέση εργασίας, ψευδής αυτοαπασχόληση, καμία εξασφάλιση για αυτού του ανθρώπους, κοινωνική ασφάλιση που έχει τεράστιες συνέπειες και στην ποιότητα ζωής των πολιτών η έκθεση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ε, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αλλά ε, θεωρώ ότι υποσκάπτεται από το γεγονό ότι δεν υπάρχει πολιτική ευαισθησία και αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Ο κόσμο αλλάζει, ε, αλλάζει το κλίμα και υπάρχει πλήρη αποσύνδεση μεταξύ αυτών και των ευρωπαϊκών δομών και των θεσμικών οργάνων για τον τρόπο με τον οποίο θα τα αντιμετωπίσουμε. Ακόμα και ένα κράτο μέλο προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει, ε, του δεσμεύουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στις συνθήκες μας. Τα προβλήματα αυτά δεν θα λυθούν με τεχνικές λύσεις και εμβαλωματικά ε, μέτρα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να σταματήσουμε τον φιλελευθερισμό. Συνεχίζουμε. Ε. σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστάσεων της Κομισιόν κατά χώρα όμω βάσει οδηγιών τη ευρωπαϊκή ένωση τα όρια συνταξιοδότηση αυξάνονται περαιτέρω η κοινωνική ασφάλιση ιδιωτικοποιείται σαν αποτέλεσμα του ΠΕΠ, μειώνονται οι συντάξει, οι συλλογικέ διαπραγματεύσει διαλύονται, μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στη δράση των συνδικάτων, περιορίζεται το δικαίωμα στην απεργία, απελευθερώνονται οι απολύσει ο Ευρωπαϊκό πυλώνα δικαιωμάτων η λογική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο, έχουν σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση του συνόλου των δικαιωμάτων προ τα κάτω ιδιαίτερα για νέου, ιδιαίτερα για γυναίκε. ο μέσο μισθό υποχωρεί αυτό δείχνουν τα στοιχεία. στην ευρωπαϊκή ένωση ζουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια φτωχοί 20 εκατομμύρια άνεργοι 5 εκατομμύρια άστεγοι ταυτόχρονα οι θέσει εργασία που δημιουργούνται το ένα τρίτο του είναι ελαστική απασχόληση που δεν καλύπτουν τι βασικέ ανάγκε. αυτά είναι τα αποτελέσματα των αντεργατικών κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής ένωσης εξειδικευμένα από τις κυβερνήσεις σε κάθε χώρα με στόχο να στηριχτεί η κερδοφορία των ομίλων καθώς στο βάθος διακρίνεται νέα καπιταλιστική κρίση. οι εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει συλλογικά οργανωμένα να απαντήσουν μέσα από τα ταξικά του συνδικάτα βάζοντα την ημερήσια διάταξη την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματά του για μόνιμη σταθερή δουλειά συλλογικέ συμβάσει που εξασφαλίζουν αξιοπρεπεί μισθού και όρια και όρου εργασία δωρεάν περίθαλψη και ασφάλιση με ευθύνη του κράτου. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ πέρα η γενική συζήτηση. Κυρία Τάισεν, έχετε εκ νέου τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία ε, Ισηγητά, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτήν την επικοδομητική συζήτηση. Σημείωσα τι θέσει σα, τι ανησυχίε σα, τα σχόλιά σα και θα φροντίσω να τα διαβιβάσω και στου διαδόχου μου. Επαναβεβαιώθηκε λοιπόν η δέσμευσή μα για μια κοινωνική Ευρώπη και για την κοινωνική οικονομία της αγοράς τις δύο όψεις δηλαδή του ίδιου νομίσματος που ενισχύουν η μία την άλλη. Η αρχή αυτή πρέπει να κατευθύνει όλο μας το έργο από εδώ και μπρος. Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε πρόκειται για την τελευταία μου συζήτηση εδώ ως ε, Επίτροπος και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία. Βεβαίως ε, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Ήμουν και εγώ ευρωβουλευτή για πάνω από 20 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια συνεργαστήκαμε επικοδομητικά, φιλικά και πάντα είχαμε κατά νου τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Τους τελευταίους μήνες λαμβάνω συγχαρητήρια για το ότι η Ευρώπη έχει γίνει πιο κοινωνική και έχει έρθει πιο κοντά στο λαό. Πάντα απαντάω ότι αυτά τα συγχαρητήρια αφορούν άλλους και θα ήθελα να τα διαβιβάσω σε εσά γιατί τα καλά αποτελέσματα είναι ο καρπός του ειλικρινούς διοργανικού διαλόγου. Τα αποτελέσματα τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στην πολιτική. έχουμε αποτελέσματα δηλαδή και να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται μια δυναμική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και μετά από 30 χρόνια στην πολιτική μπορώ να πω πως είμαι υπερήφανη για τα όσα έχω πετύχει και έχω πολλές ελπίδες για τα όσα ακολουθούν, αλλά μην με παρεξηγήσετε. Υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις μπροστά μας. Τώρα το συζητάγαμε. Και η δίκαιη μετάβαση δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αυτομάτως. Αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές της νέας Προέδρου, της ε, κυρίας Φόντερ Λάιν, δείχνουν πως η διαδοχή μας θα οικοδομήσουν σε αυτά τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί με βάση τις κοινέ μας αξίες. Σας εύχομαι λοιπόν μια επικοδομητική θητεία και πάντα θα είμαι στο πλευρό σας για μια κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ακούσατε το χειροκρότημα. Ε, το κοινοβούλιο σας ευχαριστεί. Ε, για την συνεργασία και προσβλέπει στη μελλοντική συνεργασία. Τελειώνει η συζήτηση για την απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ με την εισηγήτρια την κυρία Τόμ. Έχετε και πάλι το λόγο, παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ. Για το ίδιο θέμα, νομίζω. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για την πολύ γόνιμη συζήτηση. Ένιωσα πολύ ευχάριστα όταν άκουσα τις ευχαριστίες των σκιωδών εισηγητών για το εξαιρετικό μου έργο. Το ανταποδίδω λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ τους σκιώδεις εισηγητές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και ευχαριστώ και την Επίτροπο Τέισεν γιατί πραγματικά έκανε μια πολύ θετική μεταστροφή προς τα κοινωνικά ζητήματα και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Μερικοί είπαν ότι θα καταψηφίσουν την έκθεση είτε γιατί είναι υπερηρεσιόδοξη και πολύ φιλόδοξη, είτε γιατί δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Αλλά ε, να έχετε κατά νου ότι ό,τι και αν κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα συμβιβασμό, συμβαστική λύση. Ε, δεν νοείται συμβαστική λύση που ικανοποιεί τους πάντες. Αυτό αποκλείεται. Όταν, όσο εκπονούσα την έκθεση, στάθηκα σε κάποια λέξη κλειδιά. Την αγορά εργασίας, την ανεργία, τι γυναίκε στην αγορά εργασίας, ε, τα παιδιά, ε, ομάδες με αναπηρίες, ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, δικαιώματα ε, ε, εργαζομένων σε online πλατφόρμες, ε, μείωση της φτώχειας, υγειονομική περίθαλψη, ψυχική υγεία. Μου είπε κάποιος χθε μέσα χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι η έκθεσή σου. Όλα τα καλά απέναντι σε όλα τα αρνητικά. Όντω, συμφωνώ. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ευχολόγιο. Αλλά είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που κάνει ουσιαστικά έναν απολογισμό των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Κάντε μια προσπάθεια και λύσετε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε εγκαίρως ακριβώς την ώρα μας τη συζήτηση. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Θα ακολουθήσουν σε 10 λεπτά οι ψηφοφορίες στις 11.30 ακριβώς και μην ξεχνάτε τις κάρτες ψηφοφορίες. Ευχαριστώ.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Μέρα κατά της θανατικής ποινής. Σε έναν κόσμο στον οποίο οι αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικοποιούνται. Η θανατική ποινή είναι προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία περίπτωση. Φέτος τιμούμε ιδιαίτερος τα παιδιά, οι γονείς των οποίων καταδικάστηκαν σε θάνατο. Είμαι πεπισμένος πως ο θάνατος που επιβάλλει το κράτος δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματική δικαιοσύνη. Και ε, πρέπει επίσης να σκεφτούμε τα ψυχολογικά τραύματα που υφίστανται τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό τώρα περισσότερο από ποτέ το κοινοβούλιο μας ε, είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως ορίζουν και οι συνθήκες μας. Θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να έρθει πιο κοντά η μέρα κατά την οποία όλες οι χώρες θα έχουν καταργήσει την θανατική ποινή. Το οφείλουμε στι μελλοντικέ γενιές και σε εμάς τους ίδιους. Και είμαι σίγουρος πως αυτό είναι και το αίσθημα όλου του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στις σημερινές ψηφοφορίες και αρχίζουμε με το αίτημα επίγουσας διαδικασίας που έχει ζητήσει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Θέλει κανείς να μιλήσει υπέρ του αιτήματος αυτού. Όχι. Εναντίον ούτε. Η ψήφη υπέρ παρακαλώ του αιτήματο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στις εκθέσεις. Έκθεση Λόπεθ Αγγιλάρ. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας. Με ονομαστική κλίση, μία ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προτιμούμε, ε, ε, συγγνώμη, προχωρούμε στην έκθεση Howard, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 4 κάθετος 2019. Τροπολογίες 1 έως 11 και 13 έως 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Και τώρα η τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια το ψήφισμα στο σύνολό του και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία ε, του Περάινεν, εξ ονόματος ε, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλι υιοθέτησε τροπολογία στη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διαθροπτικού προπολογισμού υπαριθμών 4 του Γενικού Προπολογισμού για το 2019. Λαμβάνω υπόψη τι ε, διαφορέ, σημειώνω τι διαφορέ απόψε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμό 4 του 2019 που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω εκ τούτου και ω ε, εκπρόσωπο τη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμφωνώ ε, να συγκροτηθεί η διαδικασία συνδιαλλαγή όπως προβλέπει το, η παράγραφος Γ του άρθρου 341 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Οπότε, σας ευχαριστώ. Θα συγκληθεί η Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Περνάμε τώρα στη δεύτερη έκθεση του κυρίου Χαόρθ με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού για δραστικές ουσίες. Η ψηφοφορία γίνεται ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία για αντίρρηση βάσει του άρθρου 112 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή. Τρίτη αντίρρηση. Για τον αραβόσιτο. Ονομαστικά και αυτή άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη αντίρρηση για την γενετικώ τροπημένη σόγια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και η τελευταία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το γενετικό τροποποιημένο ραβό στο η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα, την ψηφοφορία ε, ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων για την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κανένα πρόβλημα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ίδια διαφορά με την πρώτη ψηφοφορία, αλλά αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, καμία αντίρρηση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 ή μάλλον συγγνώμη, τροπολογία 14 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία... Ε, όχι, δεν πρόκειται. Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε πάντα ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα. Η ίδια διαφορά ισχύει και εδώ. Αλλά αν θέλετε και τρίτη φορά, καλός ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία για τη 14. Τροπολογία 14. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχω καλή ορατότητα από εδώ πέρα για το αποτέλεσμα. 3. Τροπολογία. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες τώρα 1 και 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα εγώ προτιμώ να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, αλλά με μικρή διαφορά. Απορρίπτεται πάντως. Ψηφίζουμε τώρα το αρχικό κείμενο της παραγράφου 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε καλό κακό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Όντως εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 21, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλό, σας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11D με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν συμμετείχαν και πολλοί στην ψηφοφορία. Επανάληψη. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τροπολογία 6. ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται και σας ευχαριστώ Περνάμε τώρα στο πι δελτα πι. Ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 4, το αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία. Με αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Έγκρινεται. Και μέρος δεύτερο πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 με ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 5 του αρχικού κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία Πέρας. Ε, εγκρίνεται. 14 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας απορριφτεται 7 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 8 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. 19, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. πέρας απορρίπτεται 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 16 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται και ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Τόμ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1 σε 3 μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος τρίτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα της Επιτροπής Απασχόλησης στο σύνολό της. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε σε λίγο στις επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ, ε, βγείτε ήσυχα από την αίθουσα. Παρακαλώ, αν δεν θέλετε να μείνετε για επεξήγηση ψήφου ή να ακούσετε τις επεξήγησεις ψήφου, βγείτε από την αίθουσα. Ευχαριστώ. out of the room if you don't want to take part. The others would like to continue. Παρακαλώ δεν λάβετε μέρος ε, στις επεξηγήσεις ψήφου. Ε, βγείτε από την αίθουσα γιατί οι υπόλοιποι θα ήθελαν να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, όσοι έχουν παραμείνει στην αίθουσα, τουλάχιστον να κρατήσουν σε χαμηλού τόνους συνομιλίε γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Ο κύριος Χέρμαν Τέρτ, αν είναι παρόν, θα λάβει το λόγο για αιτιολόγηση ψήφου. Από εδώ δεν τον βλέπω, δεν ξέρω που είναι. Αφορά την αντίρρηση δυνάμει του άρθρου 112 για τον γενετικό στροποποιημένο αραβόσιτο. Ο κύριος Στέρτς είναι παρόν. Όχι, αλλά είναι ο κύριος Πόλτσακ που έχει τη δεύτερη αιτιολόγηση ψήφου. Για ένα λεπτό κύριε Πόλτσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ε, στο θέμα αυτό δεν ήξερα τι να ψηφίσω. Ε, τελικά αποφάσισα να καταψηφίσω. Δεν συνηθίζω να είμαι γενικά κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ε, αλλά ε, ε, αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να τηρούμε πολύ αυστηρά κριτήρια για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. εδώ δεν χωρούν αμφιβολίες και αμφιτέλαντευσης. Αν αρχίσουμε να επιτρέπουμε την αγορά, μάλλον την πρόσβαση σε αγορά για προϊόντα τρίτων χωρών, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να είναι ασφαλή και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μου φαίνεται σωστό να εισάγουμε αραβόσιτο από τόσο μακριά από την Νότια Αμερική ε, και να είναι προβληματική αυτή η εισαγωγή και η χρήση. Uh, Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στην αντίρρηση βάση του άρθρου 112 σχετικά με τη γενετικά τροποποιημένη σόγια. Η κυρία Κιλάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταψηφίζω και τις τρεις αντιρρήσεις ε, για σήμερα σχετικά με την έγκριση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για διάφορους λόγους. Οι συστηματικές αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα δεν βασίζονται σε τεχνικές γνώσεις, αλλά σε συναισθήματα, προκαταλήψεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες για την ε, υποβολή της αίτηση. Έκανε αξιολόγηση κινδύνου η ΕΦΣΑ και κατέληξε ότι είναι τόσο ασφαλή τα προϊόντα όσο και τα συμβατικά. Υπάρχει συνένεση των επιστημόνων σχετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και το κοινοβούλιο μας δεν μπορεί να στηρίξει αντιρρήσεις που στερούνται κάθε επιστημονικής βάσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλτσακ είναι και πάλι ε, ο μιλητής για τη ολογήση ψήφου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ προηγουμένως ε, σας ανέφερα τη θέση μου για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Οι κανόνες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηροί και επιστημονικά τεκμηριωμένοι. Γι' αυτό καταψήφισα την αντίληση για τη σόγια. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, γίνεται η καλλιέργεια αυτών των προϊόντων σε τρίτες χώρες. Για παράδειγμα στη Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει μια χώρα που εξάγει μαζικά τέτοια προϊόντα. Και εμείς έχουμε μεγάλη ανάγκη από πρωτεϊνούχες ε, καλλιέργειες και ε, η συνέπεια αυτής της μεγάλης ζήτησης είναι η αποψήλωση ε, του Αμαζονίου για να γίνουν μόνο καλλιέργειες. Είναι λοιπόν ανάγκη να τηρήσουμε αυστηρέ προδιαγραφέ για τους γενετικώ τροπημένου οργανισμούς και αν τους δεχτούμε μόνο υπό ώρες και να είναι σαφής ε, η θέση μας χωρίς διπλά μέτρα και σταθμά. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ε, ξένη παρέμβαση σε δημοκρατικές εκλογικέ διαδικασίε. Η κυρία Στρουγκάριου είναι η πρώτη που θα κάνει αιτιολόγηση ψήφου για το ψήφισμα αυτό. Είστε εδώ, ναι. Θα συνεχίσω στα ρουμανικά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις παραπληροφόρησης από hacker ε, Ρώσους. Ε, μάλιστα τα κρούσματα αυτά έχουν διπλασιαστεί φέτος σε σχέση με το 2018. Έχουν, έχουμε εντοπίσει πάνω από χίλιες τέτοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένη και πολύ στοχευμένη αυτή η παραπληροφόρηση. Το μήνα αυτό ένας Ρουμάνος δημοσιογράφος ανακάλυψε ότι ένα κανάλι με δελτίο ε, με ειδήσεων είχε πάνω από πέντε ψεύτικους, οργανισ... Ε, ψεύτικους λογαριασμούς στο ίντερνετ η, Μόσχα χρησιμοποιεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Εμεί λοιπόν θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειε μα για να αντικρούσουμε τέτοια παραπληροφόρηση. Και θα ήθελα να ζητήσω από το νέο υπατό εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική να γίνει η Stratcom μια μόνιμη δομή, ένα μόνιμος φορέα γιατί χρειαζόμαστε ξεκάθαρο πρόγραμμα για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση και να διαπαιδαγωγήσουμε το ευρωπαϊκό κενό. Ο κύριος Κυρία Μπομ. Σας ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ την ε, Λετωνία και βεβαίως υπερψήφισα γιατί όλη η Ευρώπη και όλα τα κράτη-μέλη που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνεχώς ε, αντιμετωπίζουν την ξένη παρέμβαση στις εκλογές. Οι Ρώσοι ανοιχτά λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν έναν ενιαίο πολιτισμικό χώρο στις γειτονικές τους χώρες και στις Βαλτικές και ήδη από το 2016 εμείς ε, ε, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και πρέπει να εργαστούμε με τρόπο ολοκληρωμένο. Και πρέπει ακριβώ να ενισχύσουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την ε, δημοκρατία και όχι μόνο κατά τις ε, χρόνιες εκλογών. Έτσι θα ενισχυθούν τα ισχυρά εθνικά ε, μημιέ κρατικά μημιέ αλλά και τα εμπορικά και τοπικά επίσης. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε άλλες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ταυτόχρονα μία διάσκεψη. Ε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε όμως, λέει η Πρόεδρος. Ε, μία φράση ακόμα, λοιπόν. Παράλληλα με την Ολομέλεια, στον οίκο της Ευρώπης υπάρχει μία διάσκεψη εγκυκλοπαίδειες εκεί εκπροσωπούνται από όλα τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει δηλαδή να δούμε το θέμα αυτό για την διατήρηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Wallace. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ το καταψήφισα γιατί είναι φάρσα αυτό. Δηλαδή υπονοεί ότι Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Βόρεια, Κορέα και Βενεζουέλα διασπείρουν παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου αναφέρεται ότι το ψήφισμα αυτό το ίδιο είναι μέρος εκστρατείας ε, παραπληροφόρησης ε, που ξεκίνησε από το ΝΑΤΟ. Δείτε τις είπα. Από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου έχουν ανατρέψει πάνω από 50 ξένες κυβερνήσεις, ε, δημοκρατικές οι περισσότερες, έχουν παρέμβει σε εκλογές 30 χωρών, έχουν αποπειραθεί να δολοφονήσουν 50 ξένους ηγέτες, έχουν ρίξει βόμβες σε 30 χώρες περίπου. Πότε θα επιβάλλουμε ε, κυρώσεις κατά της χώρας αυτής δηλαδή, ενώ επιβάλλουμε κυρώσεις κατά της Κρυμαίας, ε, Κίνας, Βενεζουέλας κτλ. Για να, για να αλλάξουν πολιτική θέση. Αυτή είναι η χειρότερη πολιτική παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Μαρία. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ καταψήφισα αυτό το κείμενο, διότι όπως είπε και ο προλαλής σας δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Υπάρχουν υπενιγμοί που συνεχίζουν αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα και όσοι είναι κατά της κυρίαρχης άποψης και των ευλογιών ε, των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς είναι απέναντι στρέφονται κατά δύο-τρία χωρών. Θυμίζω ότι στην Γαλλία εκπέμπει το Russia Today, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί παραπληροφόρηση. Η μόνη παραπληροφόρηση και λανθασμένη που είχαμε μαζικά στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, και το θυμάμαι, ήταν για τη Συρία και αυτό το... Ε, έκαναν τα κρατικά κανάλια όπου περιέφεραν ένα ψευτοδήμαρχο του Χαλεπιού που έλεγε ότι το Χαλέπι είναι χάλια και τα λοιπά και μετά δεν ήταν αυτός καν δήμαρχος και ήταν κατασκευάσματα ε, όλα αυτά. Άρα δεν ε, έχουμε να δώσουμε διδάγματα σε κανένα. Ο κύριος Χουκ, κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι σημαντική η ακαιρεότητα των εκλογών για την επιβίωση της ίδιας της δημοκρατίας. Μία έκθεση της Βρετανικής κυβέρνησης ε, λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε παρέμβαση ξένη ε, στο δημοψήφισμα του 2016. Ρώσικα μέσα ε, έκαναν πληροφόρηση και διέσπηραν ψευδείς ειδήσει. Και ε, η χρηματοδότηση των κομμάτων χωλαίνει πάρα πολύ νομοθετικά στη χώρα μου και ιδιώτες και εταιρείε μπορούν να δίνουν χρήματα ε, και είναι πραγματικά γνωστό. Δεν υπάρχει τρόπος να ε, ελέγξει κανείς αν προέρχονται τα χρήματα από ξένη χώρα, πόσο μάλλον από ξένη κυβέρνηση. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που τα ελέγχουν και πολλοί από αυτούς δεν ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι θέμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε για να το λύσουμε. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ρόουετ. Ε, είχαμε τραγικά συμβάντα αυτή την εβδομάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός των συνόρων μας. Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των απόψεων και της, της, ε, της, ε, των ειδήσεων και της πραγματικότητας. Τα αδιανόητα γίνονται πια πίστευτα και λαμβάνουν χώρα. Και μάλιστα μερικές, κάποια παραπληροφόρηση ξεκινάει από τις δικές μας ολιγαρχικές ελίτ. Μερικές βέβαια προέρχονται από εξωτερικές πηγές. χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρούς έγκυρους κανονισμούς για την χρηματοδότηση των, ε, εκλογικών, ε, των εκλογών, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα αίτια, την αύξηση των ανισοτήτων, ε, την απαράδεκτη, τον απαράδεκτο πλουτισμό των λίγων. Επίσης χρειαζόμαστε και παγκόσμια ισχυρά μέσα για να καταπολεμήσουμε την ξένη παρέμβαση. Υπερψήφισα ε, το ψήφισμα γιατί χρησιμοποιούμε μια πολιτική φιλία. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να διατρανώσουν τη φωνή τους και να ακουστεί η φωνή της ενότητας και της διαφορετικότητας σε όλες τις συζητήσεις μεταξύ αδερφών ε, και στην Υπηρώ μας και διεπιρωτικά. Αλλά θα πρέπει να μειώσουμε την ένταση των φωνών, των επιθετικών φωνών που δυστυχώς ακούγονται πολύ έντονα. Ο κύριος Μωράς, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Δεν θα πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί ως προς το θέμα της ε, ξένης παρέμβασης στην ακαιρεότητα των εκλογικών διαδικασιών. Και μάλιστα ζητήσαμε τη σύσταση ειδική Εξεταστικής Επιτροπής και οριακά ε, καταρρίφθηκε αυτό το αίτημα. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί οι συνάδελφοι μίλησαν για έλλειψη τεκμηρίων. Μα ακριβώ αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να εξασφαλίσουμε στοιχεία, αποδείξεις, ότι, ώστε οι δράσεις μας να είναι τεκμηριωμένες, και να προστατεύσουμε τις εκλογές μας και τη δημοκρατική βούληση των λαών μας και στα κράτη-μέλη αλλά και σε ε, εκλογικέ διαδικασίε αλλού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, δεδομένη τη έξαρση τη παραπληροφόρηση, τη εκλογική απάτη και τη ξένη παρέμβαση στι εκλογικέ διαδικασίε πολλών χωρών μελών. Και παρόλο που τελικά δεν θα καταφέρουμε να στήσουμε αυτή την ειδική εξεταστική επιτροπή, α φροντίσουμε τουλάχιστον ώστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι επιτροπέ ΛΥΜΠΕ και να το θέμα αυτό να ε, δώσουν μια συνέχεια και να μην είμαστε συγκαταβατικοί και να προστατεύσουμε τις εκλογές μας. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα καλά τους δύο τελευταίους ομιλητές. Παρακαλώ είτε να μιλήσετε πιο δυνατά ή τεχνική να ανεβάσουν λίγο τα μικρόφωνα. Περνάμε άρα στον επόμενο ομιλητή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφιζα, υπερψήφισα το ψήφισμα, αλλά θα ήθελα να πω κάτι στους συναδέλφους. Όταν μιλάμε για ξένη παρέμβαση πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Να μην στοχεύουμε άτομα. Πρέπει να στοχεύουμε κράτη και άλλους δρόντες από τρίτες χώρες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε ένα κλίμα αυτή τη στιγμή δυσανεξίας στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξένος στην χώρα μου, στη χώρα την οποία εκπροσωπώ εδώ μέσα. Όλοι ξένοι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Ε, καμιά φορά ο όρος αυτός είναι αρνητικός. Ε, δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε έτσι εύκολα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επεκταθεί το δικαίωμα ψήφου σε όλους όσους κατοικούν στην Σκοτία. μοιραστούμε λοιπόν τις δημοκρατικές μας αξίες ε, για να μπορούν να ψηφίζουν όλοι είτε είναι ξένοι είτε όχι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε την ξένη παρέμβαση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ψήφισμα για την ξένη παρέμβαση. Το σημαντικό λοιπόν είναι το ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη οικονομική στήριξη από την Stratcom. Η ομάδα αυτή ασχολείται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Fox. Εγώ το καταψήφισα αυτό γιατί τι λέει και σβήνει το μικρόφωνο. Τι λέει για τους ψηφοφόρους, ήσασταν χαζοί, δεν μπορείτε να αποφασίζετε και δεν ξέρετε τι κάνετε. Όσον αφορά τα... την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσει ακούγονται αρκετά εδώ πέρα πράγματα, συκοφαντικά μάλιστα. Να σας πω το εξής, οι ψηφοφόροι του Brexit δεν ψήφισαν λόγω Facebook ή Ρώσων πρακτόρων, αλλά επειδή πιστεύουμε στην κυριαρχία. Θέλω να προειδοποιήσω τους ε, φίλους μας ε, στην Ευρώπη για κάτι. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει στι εθνικέ εκλογέ όταν γίνονται δημοψίσματα. Ιρλανδία, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο μα λένε «Ε, ψηφίσατε λάθο. Α, ξαναψηφίστε και ξαναψηφίστε μέχρι να ψηφίσετε αυτό που θέμε. Και το ψήφισμα αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να λογοκρίνει το τι διαβάζουμε. Το καταψήφισα γιατί είναι επίθεση κατά των ψηφοφόρων. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Σντάνοκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ το καταψήφισα αυτό. Πρέπει απλά να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά όχι με τα μέσα που προτείνονται εδώ. Λέει εδώ να αναβαθμιστεί η Stratcom σε μόνιμη ε, δομή με μεγαλύτερη χρηματοδότηση και ταυτόχρονα βρίσκουμε την ε, δικαιολογία ότι υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις παραπληροφόρησης το 19. Ο λόγος όμως είναι ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού και όχι το αντίστροφο. Δηλαδή η ζήτηση δημιούργησε την προσφορά. Όσον αφορά δε τους συνδρομητές της ε, Stratcom και αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα Αναφέρθηκε παραδείγματο χάρη ένα ρεπορτάζ της ρωσικής ε, τηλεόρασης ε, με ένα ζώο ε, το οποίο όμως πρόκειται για ένα περιστατικό στην δανέζικη τηλεόραση. Δηλαδή οποιαδήποτε κριτική εδώ πέρα την βαφτίζουμε παραπληροφόρηση. Εκεί πάντα εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ. Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, εγώ στήριξα το ψήφισμα αυτό Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει διάφορα συμβάντα τέτοιων παρεμβάσεων και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ αλλά το θέμα δεν είναι πάντα εξωτερικό υπάρχει χρηματοδότηση εντός της Ευρώπης ε, που στοχεύει στην αλλαγή της γνώμης ανθρώπων που θα ήθελαν να να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Το βλέπουμε αυτό στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, οι πράσινοι και άλλοι. Υπερασπίζονται εγκληματίες ε, υπό την αιγίδα της Επιτροπής του Ελσίνκη. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και είμαι κατά. Ο κύριος Πόλτσακ, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα το συγκεκριμένο ψήφισμα παρά το γεγονός ότι ε, έχει και κάποια επίμαχα σημεία. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχουν απόπειρες ε, τρίτων χωρών να ε, παρέμβουν και να επηρεάσουν τις εκλογές στην Ευρώπη, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές εκλογές είτε είναι εθνικές. Εγώ εκτιμώ πολύ ε, την Τζέσικα Όντων, μία ε, δημοσιογράφο που έχει τεκμηριώσει ε, ότι στην Αγία Πετρούπολη υπάρχει πραγματικά εκτροφή τρόλ κανονική και οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη στιγμή διεξάγουν και δικαστικές έρευνες για να δούμε αν υπάρχει πραγματικά τέτοια παρέμβαση και ποια είναι και τι συμβαίνει θα πρέπει οπωσδήποτε να σπάσουμε, να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα. Επόμενος ομιλητή είναι ο συνάδελφο Αουστρεβίτσιος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έμεινα άναυδο, όπως και εσεί, όταν μάθαμε ότι υπάρχει η P2Day, μια ψεύτικη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Stratcom διαπίστωσε ότι αυτό απορρέει από το Russia Today, αυτό το κανάλι προπαγάνδας του Κρεμλίνου. Δεν το βλέπετε αυτό παντού. Θα πρέπει να αυξήσουμε την αθεκτικότητα των πολιτών μας και τη δυνατότητά τους να διακρίνουν τις πραγματικές από τις ψευδείς ειδήσει. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, ε, την Task Force Stratcom για την Ανατολική γειτονία. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την αγωγή του πολίτου και τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης ε, των πολιτών ε, για θέματα τύπου. Θέλουμε να δοθεί περισσότερη διεθνής και ευρωπαϊκή προσοχή σε αυτό και ε, μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για τις ε, δραστηριότητες που προανέφερα. Επίσης, ο επόμενος υπότος εκπρόσωπος θα πρέπει να κάνει την καταπολέμηση της ε, παραπληροφόρησης ουσιαστικό στοιχείο πολιτικής και μάλιστα της εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Επόμενες επεξηγήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο τώρα και θα αρχίσουμε από την κυρία Στρουγκάριου. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί θα πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στο Συμβούλιο Νόψη και των συζητήσεων της επόμενης εβδομάδας. Και παρόλα αυτά εξεπλάγει πάρα πολύ βλέποντας ότι παρόλο που το υποστήριξαν αυτό το ψήφισμα οι τέσσερις μεγάλες πολιτικές ομάδες δεν υπήρχε ούτε λέξη για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, το μέσο για τα δικαιώματα και τις αξίες. Και δεν γίνεται πουθενά λόγος για την κοινωνία των πολιτών. Παραδοσιακά το κοινοβούλιο μας ήταν υποστηρικτής της κοινωνίας των πολιτών και χρειάζονται ε, οι πολίτες ένα μέσο για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση ε, εν και τη συζήτηση τη άλλη εβδομάδα. Περιορίζεται ο χώρο όπου μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών ε, σε χώρε όπω είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, ακόμα και η δική μου χώρα η Ρουμανία. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Γερούν Λέναρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα μας εξέπληξε ε, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ε, παραμένουν 300 ε, δισεκατομμύρια αδιάθετα. Ε, είναι τα δύο τρίτα, μάλλον διπλάσιος, σχεδόν τριπλάσιος ο προϋπολογισμός και θέλουμε να αυξήσουμε και παραπάνω. Βέβαια έχουμε το Brexit, αλλά το κόμμα μου, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα τη Ολλανδία κοιτάει πρώτα τι δαπάνε και όχι ότι μα λείπουν έσοδα. Πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίε. Οι νέε προτεραιότητε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο να πά να κρεμά και εσύ τη βαλίτσα σου, το δικό σου project. Ε, θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στη διαχείρισή μας και να μην κάνουμε πολιτικά δωράκια που θα πρέπει να πληρώνουν κάποιοι άλλοι πολίτες. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί και φιδωλοί με τα χρήματα. Ε, αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και το κόμμα μου το ΣΕΔΕΑ καταψηφίζει. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον Λέσσεκ Μίλλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε υπερψήφισα το ψήφισμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε δύο πράγματα. Καταρχήν, ε, το τοπίο για τον Brexit είναι ακόμη αβέβαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να έχει ένα plan B. Ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρίς συμφωνία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον ε, προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, εκταμίευση των κονδυλίων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δικαιούχους και για τους Πολωνούς φυσικά επικούς ε, και κυρίως τους ψηφοφόρους μου στα Βιλοπόλσκα που με με την ψήφο τους. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση του στήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την, ε, μετά την των διορθώσεων και των επιστροφών θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε νέους ιδιοσπόρους, για παράδειγμα τον ψηφια το ψηφιακό φόρο. Θα πρέπει να φορολογήσουμε τους ψηφιακούς κολοσσούς, τις μεγάλες τεχνολογικές ε, εταιρείες. Αλλά ε, και τι υπόλοιπε εταιρείε που παρόλο που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίζουν εκεί δεν ε, ε, πληρώνουν φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι έδρες τους βρίσκονται εκτός τη της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη ξέχασα να κοιτάξω το χρονόμετρο. Δικό μου λάθος και έτσι μιλήσατε λίγο παραπάνω. Ρόρι Πάλμερ. Ο, δεν θέλει το λόγο. Οπότε... Το λόγο έχει η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματός μας για το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο παρά τις αμφιβολίες που είχα. Ε, και ο κύριος Λένερς είπε ότι είχε αμφιβολίες εγώ τελικά παρά τις αφιβολίες μου υπερψήφισα γιατί καλό θα ήταν να απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταλήξουμε το συντομότερο σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα στον προπολογισμό μα και να χρηματοδοτηθούν σημαντικά προγράμματα όπω το Έρασμο, το Ορίζον Ευρώπη. Επίση, να χρηματοδοτήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική, την πολιτική συνοχή. Και είναι σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο αλλά και η συζήτηση για τους ίδιους πόρους είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλούσε για 11, εμείς για 11,3, για ένα μάλλον, και εμείς για 1,3. Νομίζω ότι είναι πιο σωστή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Μπρέτσιονοβα, εγώ καταψήφισα το ψήφισμα αυτό γιατί ε, βρήθη ε, διατυπώσεων όπως σταθερότητα, πολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά της λείπει ένα βασικό κοινωνικό σχέδιο. Και επίσης το ψήφισμα ζητά την θέσπιση εταιρικού φόρου, του φόρου των ψηφιακών υπηρεσιών, φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, προσαρμογή του τελεστού του ΦΠΑ και το καθεξής. Αντιλαμβάνομαι ε, τις προσπάθειες των σοσιαλιστών συναδέλφων, αλλά πραγματικά με ευνηδιάζει και με εκπλήσει η θέση πολλών ευρωβουλευτών που αυτοποκαλούνται κεντροδεξί. Νομίζω ουσιαστικά το ψήφισμα συνιστά μια έκκληση για αύξηση των φόρων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαμπάσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ στήριξα το ψήφισμα αυτό το οποίο είναι μέρος της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επηρεαστούν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ. Το ψήφισμα περιέχει διάφορες θέσεις ε, που έχουμε στηρίξει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το σχέδιο δράσης για καταστάσεις ανάγκης ένα δίκτυο ασφαλείας για να υπερασπιστούμε τους δικαιούχους ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να καταστεί δυνατό να επεκταθεί το τρέχον πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γουάλλας θα ήταν ο επόμενος ομιλητής, αλλά αποχώρησε. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα. Πολιτική για την απασχόληση στην ζώνη του ευρώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Πάλμερ. Ευχαριστώ. Αναφέρω κατά λέξη. Οι εργαζόμενοι φεύγουν από εδώ και από εκεί, απολύονται με την πρώτη ευκαιρία. Είναι απαράδεκτο περιβάλλον εργασίας. Ε, τα αποτελέσματα βγήκαν και θα απεργήσουμε. Αυτά ένας εργαζόμενος στη Γουλκο, στην περιφέρειά μου, που θα απεργήσουν αύριο με το συνδικάτο τους. Η Γουλκο ήταν μια οικογενειακή εταιρεία με αξίες ε, που είχε δεσμούς με την τοπική κοινότητα. Δυστυχώς είχε απομακρυνθεί από αυτά και θα ήθελα εγώ να στηρίξω πλήρως ε, την, τους εργαζόμενους εκεί που αναλαμβάνουν δράση κατά αυτών των νέων πρακτικών που θα αναγκάσουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερο, κάτι το οποίο τους επιβλήθηκε με τρόπο άδικο. Και το συνδικάτο τους ε, και οι εργαζόμενοι έχουν την στήριξή μου. Σας ευχαριστώ η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ πέρα θα ήθελα να εξηγήσω το γιατί στήριξα αυτήν την ε, έκθεση. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές ε, προτάσεις που πρέπει να προωθηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη για να μην έχουμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών παραδείγματο χάρη πρόσβαση σε μέτρα απασχόλησης ε, για τους ε, νέους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, δυνατότητες. Αρκεί να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Μετά έχουμε το θέμα της εκπαίδευσης, αμοιβαία αναγνώρισης των προσόντων κτλ. Δεν λέω να έχουμε ευρωπαϊκό επίδομα ανεργία, αλλά συντονισμό θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ. Απήχα. Γιατί παρά το ότι θέλω να αντιμετωπιστεί η ανεργία, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι εγγυάται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ψευδής είδηση. Πάλεψαν για 7 εκατομμύρια άνθρωποι ενάντια στα αφεντικά τους και τις κυβερνήσεις. Και όμως εσείς λέτε ότι παραχωρήσατε δικαιώματα σαν ψίχουλα με έξτρα γραφειοκρατία. Και όλα αυτά που μας λέτε πώς τα ακούνε στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης που τιμώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την λιτότητα, την ανεργία και ταπείνωσε τα κράτη λέγοντας ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν την οικονομική τους πολιτική. Απήχα λοιπόν γιατί συμφωνώ με τη στήριξη των δικαιωμάτων των εργατών αλλά δεν εμπιστεύομαι τα μούτρα σας, φοβούμε και απευθύνω έκκληση στους φίλους Ευρωπαίους να μην βασίζονται στους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Και τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση ήταν ισορροπημένη και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής διάστασης και της κοινωνικής. Επίσης, ε, να προωθήσουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ε, αναγνωρίζει τη μεγάλη μεταναστευτική πίεση που νιώθουν τα κράτη-μέλη και μάλιστα είχαμε πρόσφατα δύο επίσης ισορροπημένες εκθέσεις για το θέμα αυτό. Ε, και περιλάβαμε και ε, τη μεταναστευτική πτυχή. Ε, το συγκεκριμένο όμως κείμενο δεν λαμβάνει δεόντω υπόψη την αρχή τη επικουρικότητα που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ασχοληθούν μετά του οίκου του σε εθνικό επίπεδο. γι' αυτό λοιπόν προτίμησα να κρατήσω στάση αποχής. Ευχαριστώ. Τα συνοπτικά πρακτικά, τα σημερινά και τα χτεσινά θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνόδου. Εάν δεν διαφωνείτε θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στους αρμοδίους φορείς και πρόσωπα. Διακόπτεται η Σύνοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, λίγη συνεδρίαση και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδας.